Just a quick announcement. If you have not yet... Αν δεν έχετε ακόμα συμπληρώσει τα έντυπα για την αποζημίωση, ε, πηγαίνετε να βρείτε τους οργανωτές έξω από την αίθουσα. Πρέπει να το συμπληρώσετε μέχρι τις 3, έτσι. Αν θέλετε λοιπόν να αποζημιωθείτε για την έλευσή σας εδώ, φροντίστε το τώρα. Use your please. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ αν θέλετε κάτι να πείτε. Εκτός μικροφώνου ήταν η ερώτηση, δεν την ακούσαμε στις καμπίνες. Νομίζουμε πως ναι, απαντάει η συντονίστρια. Πού είναι ο Αντώνιο. Μπορούν αργότερα να υποβάλουν, ε, Αγγέλικα, μπορεί να γίνει αργότερα υποβολή. Μπορούν να υποβάλουν τα έντυπα αποζημίωσης και αργότερα. Εκτός μικροφώνου οι παρεμβάσεις δεν ακούγονται στην, ε, στους διερμηνείς. Μέχρι τις 3.30 λοιπόν, αν θέλετε. Εδώ αλλά μπορείτε και να το στείλετε. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω, hashtag IW2 2018 Επίσης hashtag Women and Tech, Women and Media. Ονομάζομαι Sheryl Miller. Είμαι η συντονίστρια σήμερα για το θέμα που όλοι γνωρίζετε πόσο πολύ με ενδιαφέρει. Είναι το πώς θα δώσουμε περισσότερη δύναμη στις γυναίκες και στα κορίτσια στα μέσα ενημέρωσης για το μέλλον. Τώρα αυτό το να δώσω περισσότερη δύναμη, δυνατέ είμαστε, περισσότερε ευκαιρίε χρειαζόμαστε. Αυτό είναι που δεν έχουμε. Σίγουρα πάντω συμφωνώ ότι τα μέσα ενημέρωση και η πληροφορική αποτελούν και το κλειδί για το μέλλον. Οπότε εδώ το πάνελ που έχουμε σίγουρα θα συμφωνήσει μαζί μου. Είναι μεγάλη τιμή για μας που έχουμε συγκεντρώσει τόσες προσωπικότητες. Εδώ στο πάνελ τους έχουμε όλους. Εξ αριστερών μου εδώ η Σάσκια Φανούφελεν που είναι διευθύνων σύμβουλος της ε, Ericsson Bilax, Βέλγιο. Δεξιά μου την Terry Ρέντκε που είναι Ευρωβουλευτής των Πρασίνων και είναι και συγγήτρια του ψηφίσματος για την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων και για περισσότερη δύναμη στις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή. Και επίσης από την Πολωνία, την Καμπίλα Σίντορ που έχει ιδρύσει το Carlos Foundation και περιμένουμε και άλλη μια ευρωβουλευτή, την Ιθασκούν Μπιλμπάου Μπαραντίκα που θα έρθει σε λίγο. Μπορούμε όμως να αρχίσουμε, να δώσουμε το ανακτήριο λάκτισμα. Τέρι. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ στο πάνελ με εσά ω συντονιστή σαν έχετε κάνει καταπληκτική δουλειά. Χαίρομαι που ήρθατε εδώ τόσοι πολλοί για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα για να γνωριστούμε και να δικτυωθούμε, να δούμε πώς μπορούμε να προβάλλουμε το όλο θέμα περισσότερο. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια για αυτή την έκθεση, για τη δουλειά που κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα τελευταία χρόνια, ως Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων, προσπαθούμε να επισημάνουμε το θέμα αυτό και να το προβάλλουμε αφενός ε, στο πλαίσιο της ψηφιακής επανάστασης ε, και αφετέρου ε, στο θέμα της ισότητας των φύλων. Γιατί, όπως παρατηρούμε, εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα ανισότητα μεταξύ των φύλων στον τομέα των ICT, σε οποιασδήποτε συζητήσει για τον ψηφιακό κόσμο, οι γυναίκες παραμερίζονται, δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων και θέλουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για να δούμε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Με αυτή την έκθεση που έχουμε συντάξει προσπαθούμε να ε, εξετάσουμε συγκεκριμένα και αναλυτικά κάποιου τομεί τη κοινωνία και να δούμε τι βήματα πρέπει να υιοθετήσουν οι υπεύθυνοι χαρακτήρε πολιτική Να σα επισημαίνω δύο-τρία από αυτά γιατί δεν θέλω να βαρεθείτε ε, ούτε να σα κουράσω και ξέρω ότι όλες σα γνωρίζετε, και όλες σα γνωρίζετε πολλά για το θέμα. Το πρώτο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή επενδύει υψηλά ποσά ώστε να γίνει πραγματικότητα η ψηφιοποίηση. Να διαμορφώσει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι κοινωνίες μας. Αυτό φυσικά όλοι το βλέπουμε θετικά. Το ερώτημα που τίθεται στην έκθεση αυτή είναι πώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα. Λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση του φύλου ή απλά δίνουμε αυθαίρετα αυτά τα χρήματα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι αυτή η ψηφιοποίηση δεν μπορεί να αποκλεί τις γυναίκες. Αυτό για το οποίο κάνουμε έκκληση λοιπόν είναι στοχευμένες επενδύσεις σε προγράμματα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και επίσης προγράμματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η γυναική επιχειρηματικότητα. Γιατί όπω παρατηρούμε σήμερα, είναι πολύ πιο δύσκολο για τι γυναίκε σήμερα να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, να λάβουν χρηματοδότηση από την ιδιωτική αγορά. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια εξισορρόπηση ε, και με τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δοθούν χορηγίες και ευκαιρίες στις, γυναί... Ε, στις γυναίκες επιχειρηματίες. Το δεύτερο που θέλαμε να επισημάνουμε ήταν το ζήτημα της παιδείας. Εκεί δυστυχώς βλέπουμε ένα χάσμα που να διευρύνεται. Ένα χάσμα που δεν ήταν τόσο μεγάλο πριν από 30-40 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν υποεκπροσώπηση των γυναικών και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει όχι μόνο τις ψηφιακές δεξιότητες αλλά και ειδικότερα τις ψηφιακές δεξιότητες που αφορούν τις γυναίκες και τις νέες γυναίκες. Να υπάρξει δηλαδή χρηματοδότηση όχι μόνο για την ε, τυπική αλλά και για την άτυπη εκπαίδευση ώστε να υποστηριχθεί η κοινωνία των πολιτών, να υπάρξουν αυτές οι πύλες εισόδου ε, στον ψηφιακό κόσμο για τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια. Και το τελευταίο που ήθελα να αναφέρω γιατί πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους τα πράγματα, αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Ένα συγκεκριμένο στόχο για τις γυναίκες όσον αφορά τη βία, το λόγο μίσους και την παρενόχληση online. Αυτό δεν σημαίνει μόνο στον ψηφιακό κόσμο, υπάρχει φυσικά και στον εξωτερικό κόσμο. Εδώ που ζούμε, στην καθημερινή μας ζωή, θέλουμε να μεριμνήσουμε ώστε να αντιμετωπιστεί επιτέλους αυτό το ζήτημα. Γιατί σε πολλά κράτη-μέλη δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη. Έχουν ψηφιστεί οι νόμοι, αλλά δεν υπάρχει επαρκής δέσμευση, δεν υπάρχουν επαρκή κίνητρα για να γίνει κάτι για αυτή την κατάσταση συχνότατα δεν είναι εκπαιδευμένοι ε, το προσωπικό της αστυνομίας, ε, οι άνθρωποι που καλούνται να ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα, όπως θα έπρεπε και πολύ συχνά οι γυναίκες μένουν μόνες τους να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα. Ε, απειλή στον κυβερνοχώρο, παρενόχληση online και θέλουμε με αυτή την έκθεση να βεβαιωθούμε ότι αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ασκήσει πίεση στα κράτη-μέλη για να αρχίσουν να ασχολούνται με αυτό το πρόβλημα. Θέλω να τελειώσω με μια τελευταία δήλωση. Παρότι υπάρχουν όλε αυτέ οι δυσκολίε και τα προβλήματα, καθώ ε, εργαζόμουν για όλη αυτή την έκθεση, αντιλήφθηκα πόσο πολύ βοηθά όλη αυτή η διαδικασία ε, πόσο μας δίνει δύναμη, δεν θα πω δύναμη γιατί είπαμε ότι είμαστε δυνατές, πόσες δυνατότητε μα δίνει η ισότητα των φίλων και η ψηφιακή ανάπτυξη μαζί. Οπότε θέλω να τελειώσουμε ε, μια θετική χρειά. Να πω ότι ναι και οι γυναίκε έχουν να κερδίσουν πολλά, αλλά ειδικότερα όλοι οι κοινωνιακοί ψηφιακοί στο μέσο έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά, αν αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει όλου μα, χωρί αποκλεισμού. Και ελπίζω η συζήτηση που θα ακολουθήσει να είναι και επικριτική και επικοδομητική σήμερα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Αν δεν ήμασταν αισιόδοξοι, δεν θα ήμασταν εδώ, έτσι. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε αυτό το τμήμα της ε, συζήτησης, να δούμε κάποιες ε, βέλτιστες ε, πρακτικές, να ενθαρρύνουμε αυτά τα οποία λειτουργούν. Κάποιος ο οποίος έχει ενθαρρύνει την δική μου την δουλειά, γιατί μιλάμε για την ενθάρρυνση των γυναικών, η Σάσκια. Λοιπόν, στην εισαγωγή μου να καλωσορίσω τους άντρες. Σηκώστε τα χέρια σας. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται ε, φωτογραφία, οι πραγματικοί παρόντες ε, στην αίθουσα. Γιατί είδα εδώ πέρα την πρόσκληση που λέει δυνάμωση ε, γυναικών και κοριτσιών στα ΜΜΕ και στην πληροφορική. Χρειαζόμαστε όμως και την υποστήριξη των ανδρών για το θέμα αυτό. Είμαι η Σάσκια, δεν είμαι μηχανικός. Το επισημαίνω αυτό από την αρχή, γιατί ήδη εδώ και πολλά χρόνια έχω διοικητικέ θέσει ε, στον τομέα τη πληροφορική και τώρα των ε, τηλεπικοινωνιών. Γιατί εστιάζουμε πάρα πολύ στι ε, θετικέ επιστήμε, του μηχανικού και τα μαθηματικά, αλλά πάει ακόμη παραπέρα το θέμα. Και βεβαίω, για να είμαι και καλή Ευρωπαία πολίτη, πέρα από διευθύνουσα σύμβουλο τη Έριξον, συνεργάζομαι και με την, ε, το βελγικό κράτος και την Επίτροπο Γκάμπριελ για να μην μιλάμε μόνο για το ότι δεν υπάρχουν αρκετές γυναίκες ε, στον ψηφιακό κόσμο, αλλά για να κάνουμε και κάτι. Και μια που είστε όλοι οι δημοσιογράφοι, νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούσουμε κάποιους αριθμούς, να δούμε περί τίνος πρόκειται. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για το Βέλγιο, ε, που είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση, αν και τώρα προσπαθώ πολλέ πρωτοβουλίες να το προωθήσω το θέμα και να υπάρχουν πρότυπα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο σύστημα, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι νεαροί, όχι παιδιά, ε, μεταξύ 15 και 18 στις ε, περιπτώσεις αυτές ε, που ακολουθούν ε, τεχνικές κατευθύνσεις μόνο 5% ακολουθούν την, τις θετικές δέσμες και στην ανώτερη εκπαίδευση είναι 22% όμως. Αυτό δεν σημαίνει μετά βεβαίως πως είναι 22% των εργαζομένων στο ίδιο ρόλο γιατί μετά ξαναπέφτει σε κάτω από 10% γυναίκες που όντως εργάζονται σε κάποια δουλειά με τεχνική φύση. Από την άλλη γνωρίζετε, και τώρα μιλάω ως διευθύνουσα σύμβουλος, ε, γιατί ε, βλέπουμε αυτό το ζήτημα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Πρώτα απ' όλα ο κλάδος θέλει τις δεξιότητες. Αν δεν έχω το κατάλληλο προσωπικό δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. 50% του πληθυσμού mm. δεν ε, το ε, λαμβάνουμε υπόψη. Τις γυναίκες δηλαδή. Αν δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερες γυναίκες ε, συνδεδεμένες στον ψηφιακό κόσμο, ποτέ δεν θα ξαναστηθεί στα πόδια της οικονομία μας. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο θέμα φύλου. Είναι θέμα οικονομίας, επιχειρήσεων, επιτυχίας στις ευρωπαϊκές ε, χώρες. Το άλλο θέμα είναι ότι 65% των θέσεων εργασίας ε, δεν θα έχει την ίδια φύση που γνωρίζουμε σήμερα. Η δικιά μου η δουλειά το 2020 δεν θα απαιτεί τις ίδιες δεξιότητες. Αν δεν εκπαιδεύομαι κάθε μέρα σε νέες δεξιότητες, θα χάσω τη δουλειά μου τα επόμενα δύο χρόνια. Και βεβαίω ε, υπάρχει ακριβώ το ζήτημα τη ευθύνη ε, τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, όπου πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμο τον ρόλο της ε, διαβίου εκπαίδευση και εκεί πέρα ακριβώς είναι ο ρόλος μας ε, ως γυναίκες. Γιατί οι περισσότερες δουλειέ ε, των γυναικών είναι στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού, των πολίσεων και αλλού, αλλά όχι απαραίτητα με τις κατάλληλε δεξιότητες που θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια. Οπότε υπάρχει μεγάλη ευθύνη εδώ πέρα στο επίπεδο τη διοίκηση των εταιριών να γίνει διαβίω εκπαίδευση πρώτη προτεραιότητα. Αλλιώ θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα ανεργία ε, τα επόμενα χρόνια και ο μόνο αριθμό που θα πέσει θα είναι ο αριθμό των γυναικών. Γιατί ε, είναι περισσότερο σήμερα στην ε, πλευρά των υποστηρικτικών εργασιών ή πωλήσεων ή τέτοιων πραγμάτων που θα μετασχηματιστούν. Όπως είπα εγώ δεν είμαι μηχανικός, η εμπειρία μου είναι περισσότερο στο θέμα του μετασχηματισμού των εταιριών. Και αν είτε τις τεράστιες ευκαιρίες που έχουμε σήμερα, έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα τα πάντα είναι διασυνδεδεμένα. Στα μήνυε, στο, στη δικιά σας δουλειά του ο κάθε πολίτης θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό, γιατί οι πολίτες ε, έχουν περισσότερες πληροφορίες. Αν δείτε τους πολιτικούς, οι πολίτες θεωρούν ότι είναι καλύτερη πολιτική. Γι' αυτό ακριβώς ρωτάνε τι κάνουν οι πολιτικοί. Πριν πάνε στο γιατρό, πρώτα τον γκουγκλάρουν και, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή το γεγονός ότι όλα συνδέονται και όχι έχουν, όλοι έχουν περισσότερη πρόσβαση στα δεδομένα, αλλάζει τον κόσμο και χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα μπορούν να σκέφτονται. Ο ανταγωνισμός δεν προέρχεται από μέσα από τον κλάδο. Αντί λοιπόν να προσλαμβάνουμε τεχνολόγους ε, στον ε, κλάδο αυτόν, όλοι θα είναι τεχνολόγοι και οι τεχνολόγοι θα χρειάζονται παντού. Σημαίνει αυτό μηχανικούς, όχι. Χρειαζόμαστε άτομα τα οποία μπορούν να σκέφτονται πρωτότυπα, να δημιουργούν νέες υπηρεσίες, νέους ε, κλάδους. Ίσως μπορεί να είναι από τον τομέα των ασφαλιών, της αυτοκινητοβιομηχανίας, οτιδήποτε χρειάζεται η δυνατότητα να δημιουργώ νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέα χρηματοοικονομικά μοντέλα. Αναλυτέ μπορούν να διαβάζουν του αριθμού διαφορετικά. Ανθρώπου μπορούν να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω μόνο μου. Χρειάζομαι να φτιάξω μια λύση με βάση διαφορετικά συστατικά. Όλα αυτά είναι διαφορετικέ δεξιότητε και ψηφιακέ δεξιότητε. Και βεβαίω οι δεξιότητε αυτέ συχνά ε, βρίσκονται στις γυναίκες. Όχι πάντα. Ε, και είναι θα έλεγα θηλυκές δεξιότητες, όχι ότι είναι πάντα σε γυναίκες, γιατί και άντρες έχουν κάποιες θηλυκές δεξιότητες. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε ε, το σημερινό σημαντικό θέμα. Να μην περιοριστούμε λοιπόν μόνο στα ΜΜΕ και στην πληροφορική, αλλά γενικότερα στην συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία του αύριο, γιατί έτσι θα επιτύχουμε και θα επιτύχουν οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Κάποια στατιστικά στοιχεία. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εδώ και κάπως εγώ πέντε χρόνια, είχαμε κάποια στατιστικά δεδομένα που έλεγε ότι αν μπαίνανε στον χώρο της τεχνολογίας τόσο γυναίκες όσοι είναι και άντρες, χωρίς να πάρουν τη δουλειά των ανδρών, αλλά για να καλύψουν τις κενές θέσεις, τότε θα προσθέταμε 9 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή οικονομία, που είναι περίπου το ΑΕΠ της Δανίας. Πολύ σημαντικό στατιστικό στοιχείο εδώ. Και μάλιστα έρχεται πολύ σύντομα μια νέα έκθεση. Ίσως αύριο να τα ακούσετε από τον Επίτροπο Καμπρίελ. Και το άλλο που θέλω να σας πω, ότι αυτό το κενό στις δεξιότητες, να ξέρετε ότι μιλάμε για εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης που θα μείνουν κενές το 2020 αν δεν αποκτήσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται και που λείπουν. 1,5 εκατομμύριο κενές θέσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαιτία ακριβώς αυτού του προβλήματος της αναταραχής στην ε, ε, τεχνολογία, την πληροφορική κτλ. Αυτό σημαίνει ότι δεν εποφελούμε θα επαρκώς σήμερα. Θα πρέπει περισσότερες γυναίκες ε, να το τολμήσουν. Τώρα ήρθε και η Ευρωβουλευτής και θα σα την παρουσιάσω. Σάσκουν Μπιλμπάο Μπαραντίκα, Ισπανία. Ποια είναι η δικιά σας άποψη για αυτό το ζήτημα. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω. Αλλά βλέπετε σήμερα είναι η παραμονή Τη παγκόσμια ημέρας για τη γυναίκα και είχαμε ένα σωρό συνεντεύξεις και τα λοιπά. Μερικές ε, φορές λοιπόν αυτό πρέπει να το ξέρουμε ότι αυτό με καθυστέρησε. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να έρθω εδώ σε αυτό το σεμινάριο όπου συμμετέχουν επαγγελματίε του κλάδου των μέσων ενημέρωση, της δημοσιογραφίας. Όντω πρέπει να προωθήσουμε αλλαγέ στον κλάδο αυτό για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται η πληροφορία που θα κυκλοφορήσει και ο τρόπος με τον οποίο αυτή κυκλοφορεί. Βρισκόμαστε σε ένα ψηφιακό κόσμο και θα μιλήσω για το περιεχόμενο που κυκλοφορεί στα μέσα και πώς χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτουμε. Τι χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουμε να αποφεληθούμε από όλες τις ευκαιρίες που μας δίνει το δίκτυο. Για το περιεχόμενο Ποιο το κάνει το περιεχόμενο, το κάνουν πραγματικοί άνθρωποι, έτσι, εμείς. Και γι' αυτό ανταποκρίνεται και στα στερότυπα που έχουμε στη ζωή μας. Και βλέπουμε ότι το περιεχόμενο επηρεάζεται πάρα πολύ από την ιδέα που έχουμε για τους άντρες και τις γυναίκες. Και αν ε, αυτό το συνδυάσουμε και με το ποιοι χρησιμοποιούν περισσότερο το δίκτυο, διαπιστώνουμε ότι τελικά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η διαφορά αυτή μάλιστα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στις υπονάπτυξη χώρες και στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου. Και έχει να κάνει με το περιεχόμενο βεβαίως, αλλά και με τις ευκαιρίες που έχουν οι άντρες και οι γυναίκες προκειμένου να μπορέσουν να υποφεληθούν από τις δυνατότητες που δίνει το δίκτυο. Υπάρχει διαφορά στην χρήση, όπως είπαμε, που έχει να κάνει με δύο ανισότητες. Την πρόσβαση στο μέσο, στην πληροφορία, αλλά και στην ίδια την υποδομή των τηλεπικοινωνιών. Και αυτές είναι δύο αδυναμίες, οι οποίες τελικά καταδικάζουν περισσότερο τις γυναίκες στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και τις βάζουν σε μια δεύτερη κατηγορία, όσον αφορά αυτές τις τεχνολογίες που βοηθούν πάρα πολύ τη γνώση, την ανάπτυξη, την πρόσβαση σε θέσεις απασχόλησης, και με την οικονομία της γνώσης. Έτσι λοιπόν υπάρχει δυναμία στην εκπαίδευση και γι' αυτό σήμερα θα έπρεπε να δώσουμε μεγάλη σημασία στο περιεχόμενο. Όσον αφορά τα στερότυπα και την πρόσβαση ίσες ευκαιρίες στις θέσεις εξουσίας, πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Ούτε καν το περιεχόμενο λοιπόν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε αυτό που είμαστε πραγματικά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στι αναπτυσσόμενες χώρε. Οι περισσότερε γυναίκε που δουλεύουν στον κόσμο το κάνουν στην ύπεθρο. Και η έκθεσή μα προτείνει μέτρα προκειμένου να δώσουμε περισσότερη δύναμη στις γυναίκες αυτές που πλήττονται από αυτήν την μειονεξία κατά κάποιο τρόπο και να τις βοηθήσουμε να είναι περισσότερο παρούσες στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανισότητα, τη φτώχεια, την ε, δικογενειακή βία. Είναι αλήθεια ότι ο ψηφικός χώρος αλλάζει τα σύνορα, επιτρέπει περισσότερη κατάρτιση και δίνει μέσα ώστε να κυκλοφορήσει η γνώση. Γλώσσες που κυκλοφορούν περισσότερο στο δίκτυο. Αυτό γίνεται με πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό ακριβώ είναι και η ελπίδα ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες και να σταματήσει η ανισότητα στον κόσμο. Γι' αυτό και έχουμε προσθέσει κάποιες συστάσεις στην ε, έκθεση της Άγγελα Βαλίνα και τη δικιά μου και στον ΟΗΕ θα πάμε αυτό το μήνα ακριβώ για να συμμετάχουμε στην διάσκεψη που θα γίνει εκεί για το καθεστώς των γυναικών που δουλεύουν στην Ήπεθρο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι για θέματα ισότητας η λύση πρώτα απ' όλα ξεκινάει από εμάς τις ίδιες. Εμάς πρώτα απ' όλα. Και από τη στάση μας απέναντι στον κόσμο. Πρέπει να εντοπίσουμε κάθε διάκριση που υπάρχει. Να την φωνάξουμε, να την επικρίνουμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μας βοηθούν. Είναι το πρώτο βήμα, η συνειδητοποίηση και, ο εντοπισμός της ανισότητας αυτής. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από εμά. Μπορεί να ακούγεται προκλητικό, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, αν θέλετε. Δεύτερον, υπάρχει η μόρφωση και η πρόσβαση στις υποδομές. Ακόμα πολεμάμε για να καταπολεμήσουμε τον αναλφαβητισμό. Υπάρχει λοιπόν και εκεί πρόβλημα, αλλά υπάρχει και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι στόχος όλων μας και να το προσέξουμε όλος ιδιαίτερος το πώς πλήττεται το γυναικείο φύλλο απέναντι σε αυτόν το ψηφιακό στοιχείο. Και να το λάβουμε υπόψη μας στις στατιστικές μας. Πρέπει να εκτιμήσουμε και να διορθώσουμε την κατάσταση. Το διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν ώστε να δώσουμε περισσότερη δύναμη στις γυναίκες και αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν οι γυναίκες συμμετέχουν πλήρως στον παραγωγικό ιστό, εξίσου όπως και οι άντρες. Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι κάτι βασικό για να το πετύχουν. Επίσης υπάρχουν και άλλες στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν. Η ιδιοκτησία γης, η χρηματοδότηση, οι υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη και τις τηλεπικοινωνίες. Μπορεί να γίνει ένα άλμα χάρη ακριβώς αυτό το παράθυρο που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι θα αποκτήσουν περισσότερη δύναμη οι γυναίκες στον κόσμο. Χρειάζονται μια οι γυναίκες αυτές που τώρα είναι καταδικασμένες στην αφάνεια, στην περιθεριοποίηση. Θα είναι πιο εύκολο να προβληθούν εφόσον έχουν αυτό το κατάλληλο χώρο. Οι πιο αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν προχωρήσει με έναν τρόπο που δεν σταματάει πια. Είμαστε το 50% των δεξιοτήτων. Χρειάζεται διαφορετικός τρόπος διαχείρισης, επίλυσης ε, ε, κρίσεων και συγκρούσεων που τώρα επιλύονται από τους άντρες. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε. Και θα τελειώσω με τα Γυναίκες, ισότητα και τεχνολογία. Με αυτές τις τρεις λέξεις. Αυτό είναι το μέλλον. Ευχαριστώ. the key for the future, indeed. This... Δηλαδή, μέλλοντος, μάλιστα. Δεν είναι εύκολο όμως ε, γιατί το φύλλο είναι οριζόντιο θέμα, η τεχνολογία είναι οριζόντιο θέμα και ακριβώ εκεί όπου διασταυρώνονται αυτά τα θέματα πρέπει να, είσαι κανείς, πρέπει να είναι κανείς ε, πανταχού παρόν και ανα πάσα στιγμή εγώ θα ήθελα να κλωνοποιήσω αυτήν. Οπότε, μιλώντας για την αποστολή αυτή, είπα ότι θα έχουμε θετικό πνεύμα, υπογραμμίζοντας ότι στον ανεπτυγμένο κόσμο τα κορίτσια μας αποκλείονται ε, δεν ε, επιχούν ηγετικό ρόλο στην ε, ψηφιακή κοινωνία. Υπάρχει πολλή δουλειά λοιπόν στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Οπότε ας δούμε το τι κάνεις εσύ Καμίλα και να γίνει μια διάκριση επίσης μεταξύ ψηφιακής, ψηφιακού αλφαβητισμού και εμπειρογνωμοσύνη. Γιατί εντάξει όλα τα παιδιά από τεσσάρων ετών χρησιμοποιούν το iPad και το διαδίκτυο. Αλλά τι γίνεται με την τεχνική νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα, το ότι οι μηχανές πλέον μαθαίνουν και λαμβάνουν αποφάσεις αυτομάτως για εμάς, το, το που πηγαίνουμε, που θα πρέπει να πηγαίνουμε, ας πούμε, τα συστήματα πλοήγησης ή την υγεία μας. Τι κάνετε εκεί, σε αυτόν τον τομέα. Για να σας απαντήσω για αυτά που κάνω πολύ συχνά τα παιδιά, οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες αλλά δεν ξέρουν πώς να τις δημιουργήσουν. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια διάκριση μεταξύ της γνώσης της χρήσης και της γνώσης της δημιουργίας, της οικοδόμησης, κάτι καινούριο. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση από την αρχή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ Έχω μπει σε αυτό το κτίριο αρκετές φορές και μάλλον μιλάω καλά γιατί βλέπω ότι συνεχίζετε να, να με καλείτε διαρκώς. Είμαι η Καμίλα Σίντερα από την Πολωνία και πριν από περίπου 7 χρόνια αποφάσισα να υποστηρίξω τις γυναίκες. Δεν διάβασα καμία έκθεση, ούτε στατιστικά στοιχεία, ούτε στερεότυπα. Απλά σε μια συνάντηση για ειδικού ε, για ε, τεχνολογίε ε, αναδυόμενων εταιριών startups δεν υπήρχε καμία γυναίκα. Και εμένα μου αρέσει η τεχνολογία, τη λατρεύω και ήθελα να προσελκύσω περισσότερε γυναίκε στην τεχνολογία. Αλλά μα ήταν άγνωστο γιατί δεν υπήρχαν γυναίκε. Και έχω μια ερώτηση προ εσά. Πόσοι από εσά ξέρετε να κωδικοποιήσετε, να φτιάξετε κώδικα, να προγραμματίσετε έναν υπολογιστή. Σηκώστε το χέρι σας αν ξέρετε πώς να φτιάξετε λογισμικό, να προγραμματίσετε να γράψετε κώδικα. Ναι, φυσικά υπάρχει ένα άντρα. Πόσοι από εσά ξέρετε να χρησιμοποιείτε το WordPress. Πόσοι από εσά γνωρίζετε κάτι για το bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα. Α, ωραία. Ωραία, χαίρομαι λοιπόν. Ε, πριν από 7 χρόνια στη συνάντηση αυτή για τη startup οι γυναίκες ήταν κάτω από το 10% των παρισταμένων και ε, εγώ αποφάσισα ότι αυτό πρέπει να αλλάξει. Ήθελα περισσότερες γυναίκες συναδέλφους στο δωμάτιο, στην ε, αίθουσα. Και εγώ με κάτι φίλους μου ξεκινήσαμε μία οργάνωση, μάλλον όχι, οργανώσαμε ένα meet-up για γυναίκες μαζί με τις φίλες μου. Για 14 ανθρώπους στη Βαρσοβία, στην Πολωνία και μετά από μερικά χρόνια Είχαμε επεκτείνει το project αυτό σε 33 πόλεις σε 15 χώρες. Οργανώσαμε προγράμματα διδαχής σε κορίτσια στο Τόκιο, στο Μόντρεαλ, στη Ουάσιγκτον, σε ένα σωρό μέρη. Η οργανώσή μου ονομάζεται ε, Girls Carrots. Ξεκινάμε τώρα ένα ίδρυμα που ονομάζεται Carrots Foundation. Και τι κάναμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα δημιουργήσαμε κοινότητε τεχνολογικέ για τις γυναίκες, διότι χρειάζεται κανείς του συναδέλφους του, το είδο του, για να τον υποστηρίξει όταν αλλάζει κανείς καριέρα ή μαθαίνει τεχνολογίες. Το δεύτερο που κάναμε είναι διδάξαμε στις γυναίκες κώδικα, να γράφουν κώδικα, να προγραμματίζουν, γιατί αν δεν ξέρουμε πώ να γράψουμε κώδικα, μα φοβίζει ο προγραμματισμό. γιατί το θεωρούμε ότι είναι μια μαγική ικανότητα, ενώ δεν είναι. Οπότε είναι απόψε όταν πάτε σπίτια σας ε, δείτε κάποια δωρεάν μαθήματα προγραμματισμού που υπάρχουν online ε, προγράμματα συγγραφής κώδικα και θα δείτε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο δεν είναι κυπρινική επιστήμη και είναι μια επιστήμη που μπορεί να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες, περισσότερα κορίτσια και το τρίτο που κάνουμε στην οργάνωσή μου συνεργαζόμαστε με εσά, με ε, τις δημοσιογράφους και πιστεύουμε πραγματικά ότι στα meetup που κάνουμε, στα workshop, έρχονται γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν κάτι. Τι γίνεται όμως με τις γυναίκες εκείνες που φοβούνται, που δεν γνωρίζουν, που ενδιαφέρονται για κάτι άλλο. Εδώ πρέπει να δούμε τα μοντέλα, ε, ποια είναι τα υποδείγματα γυναικών ε, που επιτυγχάνουν στον τομέα της τεχνολογίας, να δείξουμε τέτοια μοντέλα για όλους και εκεί τα νεαρά κορίτσια θα μπορέσουν να βρουν το μοντέλο που τις εκπροσωπεί. Τα νεαρά αγόρια θα μπορούν να δουν, να αντιληφθούν ότι τα κορίτσια μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικού τομεί και κάποιε ενήλικες γυναίκε μάλιστα μπορεί να σκεφτούν να αλλάξουν καριέρα. Το Carrots Foundation ε, είναι ένα καλό μέρος για να αλλάξει κανείς καριέρα. Εγώ έχω δει γυναίκες να έρχονται συναντήσεις μας σε ένα workshop τριήμερο ε, στα, και είναι γύρω στα 30 αρχίζουν να γράφουν κώδικα, αντιλαμβάνονται ότι δεν χρειάζονται και μαγικές ικανότητες και αλλάζουν την καριέρα τους, βγάζουν περισσότερα χρήματα, συναντούν ένα σωρό ενδιαφέροντες ανθρώπους. Πιστεύω λοιπόν σε αυτά τα καλά παραδείγματα. Είναι καλύτερα από οποιαδήποτε πολιτική κατά την απόψη μου. Αυτό κάνουμε λοιπόν στο Ίδρυμά μας. Αλλά πέρυσι σκεφτήκαμε ότι ενδεχομένως όλες αυτές οι δεξιότητες να μην αρκούν διότι αν οι γυναίκες ξέρουν να γράψουν κώδικα, ξέρουν πώς να κατασκευάσουν τεχνητή νοημοσύνη, ε, να δημιουργήσουν νέα κρυπτονομίσματα ή να κατασκευάσουν ρομπότ. Ακόμη και τα ξέρουν όλα αυτά, αυτό δεν αρκεί γιατί πρέπει να βγουν μπροστά και να παρουσιάσουν αυτό που έχουν φτιάξει. Πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση. Πρέπει να μπορούν να μιλήσουν δημοσίως. Πρέπει να ξέρουν πώς να πουλήσουν το προϊόν, την ιδέα τους. Αυτές είναι ξεχωριστές ε, δεξιότητες και ναι, οι τεχνικές ε, δεξιότητες είναι σημαντικές αλλά και οι ήπιες, e τα soft skills αυτά είναι σημαντικά διότι αυτά είναι που θα εκτοξεύσουν τις γυναίκες σε ηγετικέ θέσεις, σε θέσεις υποδειγματικές όπου θα μπορέσουν να αποτελέσουν μοντέλα για τους άλλους και να, κάνουν μια, να ανοίξουν μια συζήτηση για το μέλλον γιατί η τεχνολογία θα είναι το μέλλον, μας αρέσει ή όχι. Θα ήθελα λοιπόν ε, ε, τελικά να σας ρωτήσω ποιοι από εσά θέλετε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες στην τεχνολογία. Σας βγάζουμε φωτογραφία, ε. Σας απαθανατίζουμε. Θα σας βρούμε μέσω τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αύριο έχουμε τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας και παρακαλούμε υποστήριξτε κάπως τις γυναίκες στο τομέα της τεχνολογίας. Πώς, πρώτα απ' όλα, μπορείτε να βρείτε κάποιες συναδέλφισές σας, φίλες σας που βρίσκονται στον τομέα, σε κάποιο τεχνολογικό τομέα που δραστηριοποιούνται εκεί και πείτε τους συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, σε θαυμάζω. Διότι πολλές φορές οι γυναίκες εγκαταλείπουν τη δουλειά τους σε ένα τεχνολογικό κλάδο, διότι διαρκώ πρέπει να αποδεικνύουν ότι ξέρουν τι κάνουν. Διαρκώ πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι αρκετά καλέ και επαρκεί. Οπότε δείξτε του λίγο θαυμασμό. Το επόμενο είναι θα μπορούσατε να ξεκινήσετε κάποια τεχνολογική δραστηριότητα εσεί και να αποτελέσετε εσεί έμπνευση για άλλου, για του συναδέλφου σα. Για τα παιδιά σα, τι ε, κόρε σα, του γιου σα, τι οικογένειέ σα. Μπορείτε να βρείτε μαθήματα online όπως σας είπα, οπότε απόψε ψάξτε να βρείτε βασικά προγράμματα προγραμματισμού ε, αυτά για χαζούλιδες όπως λέγονται for dummies ε, online, για άσχετους έτσι λέγονται. Ψάξτε να τα βρείτε λοιπόν και ελάτε στο δικό μας ε, site της carrots.org να μάθετε τι κάνουμε κι εμείς. Αν σας αρέσει τεχνολογία θα βρείτε κάτι. Αν δεν γνωρίζετε τίποτα για τεχνολογία μην ανησυχείτε. Εκεί είναι, υπάρχει ένας ασφαλής χώρος, ένας ασφαλές περιβάλλον για να μάθετε ό,τι επιθυμείτε. Ευχαριστώ. I just feel like I must be doing something. Κάτι στραβό μάλλον θα έχω κάνει, γιατί εμένα μου ζήτησαν να κάνω αυτή τη δουλειά. Ίσως δεν θυμώνω αρκετά, δεν ξέρω. Όλα Αυτά που ακούσαμε από τις ομιλήτριές μας ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Αυτοί που χρησιμοποιούν το δίκτυο με αυτούς που το φτιάχνουν, η συνάντηση στον ΟΙΕ, πώς οι γυναίκες πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία και να βγουν προς τα έξω. Θέλω να σας ενθαρρύνω, όπως κάνουμε εμείς με τις κοινότητές μας. Το Android είναι μια το IT Android είναι μια πάρα πολύ καλή πλατφόρμα για να μάθει κανείς Ψάξτε το στο Google και θα το βρείτε. MIT Inventor για το Android. Πράγματι, είναι το καλύτερο μάθημα στον κόσμο. MIT, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ερωτήσεις φαντάζομαι ότι έχετε. Να, ορίστε, είδατε ήδη. Ορίστε. Πείτε μας ε, ποια είσαστε και σε ποιον απευθύνεται η ερώτησή σας. Ευχαριστώ για όλους είναι. Είμαι Σάνεμα, είναι από την Τσεχία και είμαι συντάκτρια και σε ένα ε, συντακτική επιτροπή σε ένα παιχνίδι στην τηλεόραση. Ακούσαμε πάρα πολλά για τα μέσα ενημέρωση, την τεχνολογία. Όταν αυτά τα δύο πράγματα όμως συνδυάζονται, ακριβώς φτάνουμε σε αυτό που κάνω και εγώ στη δουλειά μου. Και αυτό ακριβώ είναι που μου άρεσε σήμερα πάρα πολύ. Γιατί για μένα είναι μια μεγάλη πλατφόρμα για νέες γυναίκες, για κορίτσια, που έτσι μπορούν να έρθουν περισσότερο σε επαφή με την τεχνολογία με ένα πιο φιλικό τρόπο. Μαθαίνουν δηλαδή μέσα από το παιχνίδι πώς να προγραμματίσουν ακόμα από μικρή ηλικία. Και είναι κάτι που δεν τους, δεν τρομάζει ακριβώς γιατί πρόκειται για ένα παιχνίδι. Και έτσι μέσα από το παιχνίδι μπορούμε να μάθουμε καλύτερα. Όσον αφορά τώρα την ε, εκπροσώπηση των γυναικών σε αυτά, είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη κίνηση φεμινισμού που και πάλι πρέπει να σας πω ότι ε, μου άρεσε πολύ. Δεν άκουσα όμως τίποτα γι' αυτό το θέμα του παιχνιδιού. Οπότε η ερώτησή μου είναι κυρίως για την έλλειψη εκπροσώπησης των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Πώς εντάσσεται το παιχνίδι σε όλα αυτά και υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε και να το στηρίξουμε περισσότερο. Για... Εντάξει, εντάξει, την καταλάβαμε την ερώτηση. Φτάνει, φτάνει, διακόπτη συντονίστρια. Καταλάβαμε. Ωραία. Ποιος θα απαντήσει. Ναι, μπορώ να προσθέσω εδώ κάτι. Είναι σημαντικό Είναι πολύ σημαντικό και οι γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, πολλές φορές ακούμε ότι άμα δεν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι εμείς που τα φτιάχνουμε πρέπει να επιλέξουμε τον τρόπο που θα τα παρουσιάσουμε στα μέσα ενημέρωσης. Να μην εμφανίζονται τόσο τεχνολογικά, σαν να πρόκειται για ένα μαγικό κόσμο που δεν καταλαβαίνει κανείς. Όχι. Δεν πρέπει να ανταποκρίνεται μόνο σε μία μικρή κοινότητα ανθρώπων. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και εμείς περισσότερο πώς θα τα παρουσιάσουμε σε μια γλώσσα έτσι πιο ανοιχτή και ξεκάθαρη. Έτσι θα βοηθήσουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν περισσότερο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και να χρησιμοποιήσουμε και τα παιχνίδια για τη δασκαλία, όπως είπατε. Συμφωνώ απόλυτα κι εγώ. Θέλω κι εγώ να προσθέσω κάτι. Εγώ δεν ε, συμμετέχω, δεν είμαι από αυτή την κοινότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά αν δείτε πώς ε, συνήθως τα παιχνίδια εμφανίζονται στην κοινωνία, πολύ συχνά οι γυναίκες εμφανίζονται σε αυτά ε, με στερεότυπα. Όταν κοιτάω γύρω μου και βλέπω τις οικογένειες, ελάχιστα εμφανίζονται καλά οι γυναίκες. Συνήθως δηλαδή δημιουργείται μια αρνητική εικόνα. Υπάρχει δηλαδή μια νοοτροπία μέσα σε αυτά που επαναλαμβάνει τα στερότυπα και πολύ σωστά τα λέτε. Τα χρησιμοποιούμε πολύ λίγο τα παιχνίδια τα ηλεκτρονικά, δυστυχώς. Και πάλι όμως επειδή είναι τα ανδροκρατικά πρότυπα που περισχύουν στα παιχνίδια αυτά. Ξέρετε ότι μέχρι τα 35 οι γυναίκες ε, ήταν οι περισσότερες. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι και εγώ συμμετέχω σε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εσείς έχω τους ε, ανιψιούς μου. Και τι διαπιστώνω τι κάνουν. Διαπιστώνω ότι πράγματι τα στερότυπα αυτά παραμένουν. Τι κάνουν οι νέοι. Ανταγωνίζονται στη βία. Ποιος θα κερδίσει στη βία. Και η συμπεριφορά τους στο παιχνίδι δεν είναι βέβαια ταυτόσιμη με την γενική συμπεριφορά. Μπορεί να μην τα ξέρω καλά τα πράγματα και εντάξει να το παραδεχτώ, αλλά δεν ξέρω καμία εταιρεία, καμία επιχείρηση που να διαλέξει γυναίκες για αυτά τα παιχνίδια. Σπάνια βλέπουμε ο πρωταγωνιστής σε αυτά τα παιχνίδια να είναι μια γυναίκα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Όταν βλέπω τα παιχνίδια, ποιοι βλέπουν αυτά τα παιχνίδια, τα παιδιά. Άρα τα παιδιά ζουν με την εκπαίδευση που παίρνουν στο σχολείο και που τους λένε πρέπει να μην είσαστε βίαιοι, να σέβεστε τις γυναίκες ε, όπως και τους άντρες. Δεν, και τι βλέπουν στα παιχνίδια, κάτι διαφορετικό. Αυτοί που κερδίζουν τη μάχη μέσα από βία συμπεριφορά βέβαια στα παιχνίδια ε, είναι άντρες. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις νέες τεχνολογίες, για τα ηλεκτρονικά αυτά παιχνίδια. Εγώ τα έχω κοιτάξει από περιέργεια και πιστεύω ότι υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο βελτίωσης. Από μικρά που είναι τα παιδιά μέχρι που μεγαλώνουν. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά ότι υπάρχουν και ηγετικές φιγούρες που είναι γυναικείες και που μπορούν να κερδίσουν. Δυστυχώς όμως και ο πόλεμος έχει αντρικό πρόσωπο. Και μέσα από τις νέες τεχνολογίες αυτό βλέπουμε. Θα πρέπει αυτό να αλλάξει, να χτιστεί η ισότητα, αλλά και μέσα από τις συμπεριφορές στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συγγνώμη, ήθελα να, να πω κάτι στα γρήγορα. Ναι, μπορείτε να το συζητήσετε προς με Απλά να πω κάτι πολύ γρήγορα. Πολλά από τα πράγματα που ακούσαμε από όλους σας Καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά ακριβώς ναι, βασίζεται σε στερεότυπα. Τα στερεότυπα ουσιαστικά εξαρτώνται από το πώς έχουν σχεδιαστεί τα games, τα παιχνίδια. Εγώ είμαι δημοσιογράφος σε αυτό το τομέα του gaming, ε, αλλά λέω όπως και άλλοι δημοσιογράφοι εδώ, ότι πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτό το τομέα. Είναι πιο ανοιχτά τα παιχνίδια, δεν κυριαρχούνται από άντρες Έχουμε πολλές ισχυρέ γυναικές προσωπικότητες μέσα στα παιχνίδια. Ε, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι ε, κλάδος αντρικός. Αυτό ήθελα να τονίσω αυτά. Ε, ξέρετε, συμφωνούμε νομίζω, ε, ε. Να προσθέσω κάτι. Η συζήτηση για το gaming είναι θέμα αντίληψης. Είναι η ίδια συζήτηση που κάνουμε για τα γυναίκες και τα ICT. Τα ICT για τα αγόρια σημαίνει ότι είναι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο πάνω σε ένα πληκτρολόγιο. Η εικόνα του κόσμου, λάθος ή σωστή, είναι αυτή που έχουμε ακούσει. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν την εικόνα. Για να σας δώσω λοιπόν ένα άλλο ξεχωριστό παράδειγμα. Αν μιλήσουμε για σοβαρό παιχνίδι, αν δούμε πώς το σοβαρό παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει να αλλάξουμε ε, τα πράγματα, να κάνουμε το μετασχηματισμό, να βοηθήσει στην εξέλιξη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ε, αν βρούμε διδάσκοντες ε, που να γνωρίζουν τον τομέα, αν το αντιμετωπίσουμε έτσι, η λέξη gaming αλλάζει μορφή. Αλλάζει η έννοια. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια παραδείγματα, κάποια μοντέλα για να αλλάξουμε. Γιατί πολλοί κόσμος, όπως ακούμε, ε, πιστεύει αυτό που ακούμε. Οπότε αυτό πρέπει να κάνουμε. Όταν μιλάμε για σοβαρά παιχνίδια, ε, βλέπουμε πολλά καλά πράγματα παγκοσμίω και πραγματικά έτσι δημιουργείται ε, πολύ, καλή, πολύ, πολύ καλά πράγματα για την οικονομία. Ωστόσο δεν ακούγεται και πολύ αστείο, έτσι δεν είναι και πολύ διασκεδαστικό. Serious gaming, σοβαρό gaming. Μήπως να οργανώσουμε αγώνες για γυναίκες. Ε, λοιπόν, να κάνουμε, ναι, να κάνουμε ένα τουρνουά για ηλεκτρονικά παιχνίδια εδώ. Ε, να παίξουμε διάφορα παιχνίδια πολεμικά και τέτοια. Ε, αλλά ξέρετε, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχουν και άλλα. Έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση και στα παιχνίδια. Κάποιο άλλο που θα ήθελε να πει κάτι ή να κάνει κάποια ερώτηση. 24 Πόλσκα. Θα ήθελα να μιλήσω ε, πολωνικά. Αφού έχω την ευκαιρία είμαι πολύ ε, χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Είμαι από την Πολωνία. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Βέλγιο. Είμαι 52 ετών και εδώ και τρει μήνε έμαθα να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο. Το οποίο μου διδάσκει η κόρη μου που είναι 13 ετών. Και ήθελα να σας πω ότι κατοικεί σε μια μεγάλη πόλη, στο Βροσλάβ, στην ε, Πολωνία μια πόλη όπου αυτή η κόρη μου δηλαδή πηγαίνει σε μαθήματα κώδικα και ήταν το μόνο κορίτσι και μαζί με 14 αγόρια στο μάθημα. Ευτυχώς ε, το μάθημα το δίδασκε μια γυναίκα και χάρη σε αυτό η κόρη μου γνωρίζει ότι μια νέα γυναίκα μπορεί να προγραμματίσει και μάλιστα καλύτερα τα αγόρια. Αυτό που με χαροποιεί σήμερα σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση είναι που βλέπω ότι εδώ Επιτέλους μιλάμε για αυτά τα νέα κορίτσια, αυτά τα καταπληκτικά νέα κορίτσια που κάθονται εδώ πίσω, στην πρώτη τελευταία σειρά, και για τα κορίτσια που είναι λιγότερο νέα, που είναι 30, 30-45 χρόνια και αυτές έχουν μια ευκαιρία την οποία μπορούν να δράξουν. Αλλά σας παρακαλώ, ας μιλήσουμε για ισορροπίες και όχι για ισότητα. Ας μιλήσουμε για ισορροπίες όσον αφορά τους άντρες και τις γυναίκες, γιατί η ανδρική ενέργεια και η γυναική ενέργεια είναι και οι δύο αναγκαίες αλληλοσυμπληρώνεται. σα το λέω εγώ, μια γυναίκα κάποιε ηλικίε. Well, we are equally old then. Ναι, έχουμε την ίδια ηλικία λοιπόν. Και εγώ κατά το ίμιση έχω πολωνικό DNA, οπότε μπράβο ε, μου λέτε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διακόψουμε εδώ τη συζήτηση, αν κατάλαβα καλά. Έχετε 10 λεπτά για καφέ Μόλις θα υπάρχει δυνατότητα λοιπόν ε, και εδώ ξέρω ότι οι συνάδελφοι θέλουν να απαντήσουν ερωτήσεις οπότε αρπάξτε τις ε, στο χολ. Ευχαριστώ πολύ στα μέλη του πάνελ που μου είχατε την τιμή να βρίσκεστε εδώ σήμερα.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

Hajar, are you here? Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουμε τώρα, θα περάσουμε στο τελευταίο πάνελ της ημέρας που είναι «Υψώνοντας τη φωνή» στο απαράδεκτο, για να αντιμετωπίσουμε το απαράδεκτο. Δυνατό θέμα, έτσι. Οπότε περιμένω να δω τι έχουν να μας πούνε όσοι βρίσκονται εδώ στο πάνελ. Πρώτα απ' όλα έχουμε την κυρία Ανιέσκα Κοστόφσκα Ραγιβίτς από την Πολωνία. Το είπα καλά, το όνομά σας το πρόφερα καλά, ρωτάει η συντονίστρια. Ο κύριος Εντουάρ Μαρτάν, εντάξει, και εσείς, η Ίγκεμπελ, που είναι από την οργάνωση Hommes και Χατιάρ Μπένι Λουτ που είναι δημοσιογράφος ιδρυτής της πλατφόρμας villain.com. Θα αρχίσουμε λοιπόν με την κυρία Κωστόφσκα Ράγεβιτς που θα μιλήσει πολωνικά, όπως έχει και το δικαίωμα. Ε? <laughs> Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω πολωνικά, οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι στην προηγούμενη συζήτηση μιλήσαμε για στερεότυπα, κλισέ, αντιλήψεις, το πώς ε, αντιλαμβανόμαστε τις γυναίκες. Η Καμίλα Σιντορόφ είχε πει το εξής όταν μπήκε σε μία συνάντηση με νεοφυείς επιχειρήσεις συνειδητοποίησε ότι μόνο άντρες υπήρχαν εκεί και αναρωτήθηκε αν είχε βρεθεί στο σωστό μέρος. Το ίδιο ισχύει και για την ε, κόρη ενός Πολωνού δημοσιογράφου που είχε πάει σε μια τάξη πολιστών και ήταν κυρίως αγόρια. και βεβαίως σε κάθε συνάντηση που πάμε στην Επιτροπή των Γυναικών πάντα υπάρχει η γυναικοκρατία όπως και εδώ πέρα σήμερα βεβαίως ε, πρέπει να απλώσουμε το χέρι στους άντρες γιατί ε, εδώ και 20 χρόνια μιλάμε σε παρόμοιες ομάδες για τα ίδια πράγματα και οι προκλήσεις παραμένουν. Παρακάτω λοιπόν βία. Ψυχολογική βία, σωματική, σεξουαλική, σεξουαλική παρενόχληση, όλα τα είδη βίας ε, θέλουμε να τα καταπολεμήσουμε. Το ίδιο και η γάμη νεαρών κοριτσιών, ε, γάμι ε, καταναγκαστική, στήρωση. Όλοι αυτοί οι τύποι βίας αφορούν ε, τις γυναίκες ως ε, θύματα, γιατί αντιλαμβάνονται τις γυναίκες με βάση κάποια στερεότυπα ως ε, κατώτερα όντα που εξαρτώνται από άλλους. Αυτό σημαίνει ότι είναι ευκολότερο να πέσουν θύματα βίας. Εντάξει, καλή η νόμη, ο ποινικό κώδικας, οι διαδικασίες και τα λοιπά αλλά δεν αρκούν. Πρέπει να προωθήσουμε την ε, ισότητα και τα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών. Η συνθήκη της ε, Κωνσταντινούπολης που έχει κυρωθεί από τα περισσότερα κράτη-μέλη προβλέπει ξεκάθαρα ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την βία. Και αυτό είναι δυνατόν εάν προωθήσουμε την ανεξαρτησία και την ισότητα των γυναικών η περισσότερες πολιτικές που εφαρμόζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνονται σε ενήλικες γυναίκες, αλλά πρέπει να δρούμε πολύ νωρίτερα. Στην ε, τελευταία συνεδρίαση του ΟΗΕ ε, πριν από ένα έτος ε, κατέστησα σαφές ότι η διάκριση εις βάρος των γυναικών είναι βαθιά ριζωμένη και ξεκινάει πολύ νωρίς όταν τα κορίτσια μπαίνουν στην εφηβεία. Είναι μια κρίσιμη φάση. Τα κορίτσια αυτά έχουν πολλές δυνατότητες μπορεί να γίνουν τραχουτίστριες ή επιστήμονες αλλά ξεκινάει μία σεξουαλικοποίηση τους ε, πολύ νωρίς ε, στο σχολείο. Ε, υπάρχει σεξουαλική βία στο σχολείο και είναι το αποτέλεσμα ακριβώς αυτής της αντιμετώπισης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα δεν ξέρω πώς θα πρέπει ακριβώς ε, να διαμορφώσουμε την πολιτική μας για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κοριτσιών και το κυριότερο πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Έχουμε νόμους, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν στην ε, πράξη. Είχαμε την ε, τελευταία συνεδρία του ΟΗΕ, του Τμήματος των Γυναικών, όπου ο Γενικός Γραμματέας είπε τα εξής μετά από πολλά χρόνια βίας κατά των γυναικών, ε, τα πάντα έχουν υποθεί, αλλά σχεδόν τίποτα δεν έχει γίνει. Οπότε η πρώτη πρόκληση για σήμερα είναι να γίνουν αυτά τα λόγια πράξη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν ε, έτσι ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος. Πέρσι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως αποκάλυψε το πολιτικό, υπήρχαν περιπτώσεις ε, πολλές σεξουαλικής παρενόχλησης. Υπήρχαν κάποια ερωτηματικά γύρω από αυτά τα σκάνδαλα. Είχαμε έρευνες ε, και πολλοί είπαν ε, ότι είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση αλλά δεν το ανέφεραν στα αρμόδια όργανα. Συμμετείχαν μόνο στην ανώνυμη έρευνα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο που πρέπει να εφαρμοστεί και είναι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης που έχει μια μεγάλη διαφορά από άλλα νομοθετήματα γιατί έχει ένα κεφάλαιο για την πρόληψη και μιλάει ακριβώς για τη σχέση καταπολέμησης της βίας και προώθησης της ισότητας. Ε, ισότητα, ίσα δικαιώματα, μείωση της βίας. Η ισότητα καθιστά τις γυναίκες ε, πιο ανθεκτικές ε, στην βία και η δυνητική επιτιθέμενοι ίσως ε, σταματήσουν πριν προχωρήσουν στην πράξη. Έτσι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας. Ευχαριστώ. Ωραία λοιπόν. Έκλεισε λοιπόν να συμμετέχουν και άντρες τώρα στη συζήτηση περισσότερων των φίλων για το θέμα αυτό που αφορά τη σεξουαλική ε, παρενόχληση, όπως επίσης και η παρουσίαση των γυναικών ως ε, παιδιών, αλλά και η παρουσίαση των κοριτσιών ως σεξουαλικών ε, αντικειμένων. Αυτό ανοίγει την πόρτα προς την παρενόχληση. Έχω λοιπόν εδώ τώρα μια παρέμβαση από τον κύριο Ματά, ο οποίος έχει ενεργά συμμετάσχει στη συζήτηση αυτή. Έχετε το λόγο. Ναι, όπως βλέπετε είμαι και έρχομαι και εγώ εδώ να μιλήσω. και είμαι μέλος της Επιτροπής ΦΑΜΑ και υπερασπίζουμε τα δικαιώματα των γυναικών ε, όπως υπερασπίζουμε τα δικαιώματα ισότητας για όλους. Για μένα δεν πρέπει να γίνεται διάκριση άντρα-γυναίκα, είναι θέμα ιδεολογίας. Ναι, στην Επιτροπή ΦΑΜΑ έχουμε όντως πλειοψηφία γυναικών, αλλά εκεί μερικές γυναίκες είναι πιο ε, συντηρητικές από κάποιους άντρες, οπότε το θέμα δεν είναι θέμα φίλου πάντα, είναι και θέμα νοοτροπίας. Είναι θέμα κοινωνία με στην οποία θέλουμε να ζούμε και να μεγαλώνουμε. Χαίρομαι ε, που άκουσα και τη συνάδελφο από το ΕΛΚ. Αυτό σημαίνει ότι θα μας είναι πιο εύκολο να πείσουμε όσου και όσε ε, εξακολουθούν να μας φέρουν μεγάλη αντίσταση σήμερα, να έχουν μεγάλες επιφυλάξεις όσον αφορά την, επικύρωση, κύρωση της, της σύμβασης Κωνσταντινούπολη, όπου συζητάμε για το πώ θα αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών. Ε, αφορά αυτή η σύμβαση και την πρόσβαση της αμβλώσης και το να διαθέτει κανείς το σώμα του όπως θέλει. Ε, εκεί έχουμε πρόβλημα, έχουμε διχογνωμία στο, και στο Κοινοβούλιο. Οπότε εκεί θα πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε όλα τα δικαιώματα των γυναικών και όχι μόνο ορισμένα για μένα. Δεν υπάρχει περιορισμό όταν αναφερόμαστε στα δικαιώματα των γυναικών. Υπάρχουν τα δικαιώματα γενικά με δέλτα κεφαλαίο. Και εμεί, όποιοι και αν είμαστε από οποιαδήποτε ε, πολιτική κατεύθυνση και αν προερχόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ναι, αυτό το δικαίωμα των γυναικών θα το συζητήσουμε και το άλλο δεν πρόκειται. Ή, ξέρω εγώ, έχουμε κάποια κόκκινη γραμμή την οποία δεν θέλουμε να υπερβούμε, διότι δεν αποτελεί κομμάτι των δικαιωμάτων που εμεί είχαμε πει ότι θα υπερασπίζουμε. Οπότε εκεί θα πρέπει να ε, αμφισβητούμε ακόμα και τα δικά μα τα πιστεύω τι συμβαίνει αυτό. Δεν μας λείπουν κείμενα, όπως είπαμε. Δεν μας λείπουν κείμενα για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης των γυναικών, ε, ε, για την ισότητα της πρόσβασης στην, ε, την ίση αμοιβή. Έχουμε πολλά ευρωπαϊκά κείμενα. Το πρόβλημα είναι η πλημελής τους η υλοποίηση, η υποκρισία από τα κράτη. Αυτό είναι κάτι βέβαιο και η δική μου χώρα, η Γαλλία, δεν είναι και η πρώτη όσον αφορά την τήρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών, ειδικότερα όσον αφορά την ισότητα της αμοιβή δεδομένων αυτών, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει και αυτή κάποια ευθύνη. Κατά την άποψή μου, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η ιεραρχή θέτει προτεραιότητες για το τι είναι σημαντικότερο για την Ευρώπη και τι είναι λιγότερο σημαντικό. Ας δούμε το χρέος των χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανελαίητα χωρίς, καμία, ε, χωρίς κανένα πρόβλημα δεν σεβάστηκε τον ελληνικό λαό και είπε εσείς δεν σέβεστε κάποια κριτήρια θα σας τιμωρήσω. Και σήμερα ο ελληνικός λαός πληρώνει ακόμα το τίμημα και Ξέρετε, το ελληνικό χρέος δεν γίνεται να εξοφληθεί. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ναι, είναι αμετάκλητη αυτή η κανόνε, έτσι έχουν τα πράγματα. Η ίδια η Κομισιόν, λοιπόν, αν είχε δείξει την ίδια αποφασιστικότητα με τα κράτη-μέλη που αρνούνται να κυρώσουν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης γιατί δεν το κάνει με τα κράτη-μέλη τα οποία δεν σέβονται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις θέσεις εργασίας, στην, ε, στις ίσες αμοιβές. Ένα σωρό περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης υπάρχουν, τις γνωρίζουμε όλοι, όλες και η Κομισιόν κάνει τα στραβά μάτια γιατί θεωρεί ότι δεν αποτελούν προτεραιότητα. δεν μπορούμε να μιλάμε για συνθήκες πρώτης κατηγορίας και δεύτερες. Η συμβίωση όλων μας είναι όλα αυτά μαζί, δεν είναι μόνο η οικονομική σύγκληση, είναι και ο σεβασμός των μειονοτήτων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων, η συμμεταχείριση, η μισθολογική πολιτική. Από τότε που εξελέγει το 2014 εγώ μάχομαι για να γίνει μια πραγματική συζήτηση και νομοθεσία για την υποχρέωση περιήση αμοιβή. Αν δείτε τους αριθμούς, τα νούμερα της Eurostat, ακόμη και σήμερα το 2018, σε αυτή την καταπληκτική τεράστια Ευρώπη που κάνει μαθήματα σε όλο τον κόσμο, έχουμε 17% διαφορά αμοιβή ε, για η ίδια εργασία. Μια γυναίκα κερδίζει 17% λιγότερο από έναν άντρα και όταν φτάνει η ηλικία τη συνταξιοδότηση η γυναίκα παίρνει 40% χαμηλότερα. Και εμεί καθόμαστε και συζητάμε αν πρέπει να ε, ε παρατείνουμε την άδεια μητρότητα ε, και υπάρχουν κάποιε προοδευτικέ δυνάμει, όχι όλοι και πάλι, και κάποιε συντηρητικέ δυνάμει και κάθε φορά λέμε ποιο θα πληρώσει ε, ε, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε υποκριτέ. Θέλουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή θέλουμε κάθε φορά να βάζουμε ένα τίμημα, μια τιμή σε κάθε πράγμα. Και εγώ ξεκινάω από την αρχή ότι η ίση μεταχείριση δεν έχει τιμή. Αλλιώ η Ευρώπη θα χάσει την πραγματική της έννοια, την ουσία της. Εκεί ακριβώς πρέπει εμείς ε, να τα συζητάμε όλα δεν μπορούμε να μην συζητάμε πράγματα, να μην επιτρέπουν να συζητηθούν πράγματα ακόμη και αυτά που μα θυμώνουν. Γιατί αν το κάνουμε, όπω κάνει συχνά η Ευρώπη, αυτό σημαίνει ότι τελικά θα συμφωνούμε σε πολύ λίγα πράγματα. Και ότι τελικά οι διακριτικέ μεταχείρισει θα συνεχίσουν για χρόνια και για χρόνια, για δεκαετίε. Και τώρα να πω και κάτι ε, για ένα θέμα που μάλλον θα μας ενώσει ελπίζω το σκάνδαλο της ε, σεξουαλικής παρενόχλησης και ορισμένα θύματα είχαν δίκιο τόλμησαν να πούν εγώ που εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ έχω υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό ξέρετε δεν άρεσε πολύ κόσμο. Με πολύ κόπο καταφέραμε να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο τον περασμένο Νοέμβριο. Έχουμε φτάσει 7 Νοεμβρίου και ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί το ψήφισμα. Γιατί? Διότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και μάλιστα το ΕΛΚ μεταξύ άλλων, το οποίο δεν θέλει να ακούει για εξωτερικούς ελεγκτές. Δεν θέλουν καν να ακούσουν λένε ας το ρυθμίσουμε μεταξύ μας. Ξέρετε τώρα πώς γίνονται τα πράγματα. Όταν δεν θέλουμε να ρυθμιστεί κάτι, λέμε ας το ρυθμίσουμε μεταξύ μα. Α τα βρούμε μεταξύ μα. Κυρίω να μην το μάθουν τα μέσα μαζικής ενημέρωση. Εγώ με τη βοηθό μου που είναι εδώ παρούσα έχουμε πει στα μέσα μαζική ενημέρωση τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποτέ δεν είπαμε ότι υπάρχει περισσότερη παρενόχληση εδώ από τέλου. Απλά είπαμε ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν περιπτώσει σεξουαλική παρενόχληση. Είναι μια μικροκοινωνία, και ε, για ποιο λόγο να είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη. Έχουμε τα καλά μας και τα κακά μας. Αλλά ευθύνη μας είναι να πούμε ότι ακόμη και αν έχουν γίνει κάποια πράγματα, πώς είναι δυνατόν τα θύματα να μην διαμαρτυρήθηκαν ποτέ στην Επιτροπή που συστάθηκε για αυτό το σκοπό. Για έναν πολύ απλό λόγο ότι η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τρεις ευρωβουλευτές από ε, εκπροσώπους ε, του προσωπικού. Ε, και συχνά είναι κοινοβουλευτικοί επιτετραμένοι αυτοί και ξέρετε, έχετε ακούσει ποτέ ένα θύμα να πάει να καταγγείλει το συνάδελφο στον ανώτερο. Ακόμη και αν το κάνει το θύμα, ξέρετε, εμεί οι Ευρωβουλευτέ μπορούμε να ξεφορτωθούμε έναν επιτετραμένο και να πούμε ότι δεν έχουμε πλέον, έχει διαραγεί η εμπιστοσύνη μα. Και εκεί έχουμε διπλή ποινή όχι μόνο το άτομο έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, αλλά διατρέχει και τον κίνδυνο να χάσει τη δουλειά του 24 ώρες μετά. Και εγώ επιμένω, πρέπει να παγιώσουμε, να προστατεύσουμε τις ε, συμβάσεις εργασίας αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να προβλέψουμε ε, τι ακριβώς σύνθεση θα έχει αυτή η Επιτροπή να την αλλάξουμε. Μπαίνουν, προσπαθούν από στη θέση των θυμάτων ε, που καλούνται να πάνε να μιλήσουν μπροστά σε άλλου βουλευτέ και να πούν τι έζησαν. Ε, ψυχολόγοι πρέπει να ακούσουν αυτού του ανθρώπου, τα θύματα, γιατροί, ε, νομικοί, όπου σε ένα περιβάλλον απόλυτη εμπιστοσύνη θα μπορεί το θύμα να πει στον εαυτό του ναι, είμαι βέβαιο, βέβαιη ότι αυτό που θα πω δεν θα βγει παρά έξω. Αλλά εντάξει, οι τρει βουλευτέ που είναι μέλη αυτή τη επιτροπή σίγουρα είναι αξιοσέβαστα άτομα και κάνουν καλά τη δουλειά του, αλλά σα το λέω ειλικρινά. Ξέρετε, δεν είναι μόνο να είναι όλο εντάξει, είναι και πώ τον βλέπουμε. Ε, έχουμε θύματα που δεν τολμάνε να πάνε σε αυτή την επιτροπή να διαμαρτυρηθούν γιατί δεν είναι βέβαιες, έτσι σκέφτονται ότι αυτά που θα πούν θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Είναι δραματικό. Πρώτο. Και δεύτερον, για να μην μονοπολώ το λόγο, πιστεύω ότι χρειάζεται εξωτερικός έλεγχος. Χρειάζεται ένα εξωτερικό μάτι. Όχι για να έρθουν να μας κρίνουν αλλά για να μας πούν, ορίστε, κοιτάξτε, αυτό γίνεται σωστά, αυτό γίνεται λιγότερο σωστά, εκεί σε αυτούς τους τομείς πρέπει να ε, γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Και τα βάζουμε αυτά στο ψήφισμά μας μετά. Αλλά για, τι, για ποιο λόγο αντιτιθέμεθα στον εξωτερικό έλεγχο. Δεν έχω λάβει κάποια απάντηση. Η απάντηση είναι πάντα ας το βρούμε μεταξύ μας. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα θύματα δεν θα τα επρασπιστούμε σωστά. Και εγώ θέλω ένα εξωτερικό μάτι, διότι εμείς εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες, την, τις κοινωνίες της Ευρώπης. Συνεπώς πρέπει να δείχνουμε διαφάνεια, να δείχνουμε ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Και μόλις πάμε και λέμε ότι δεν θέλουμε εξωτερικό έλεγχο, αυτό ε, σημαίνει κάπου ότι κάτι έχουμε να κρύψουμε. Δεν θέλω εγώ να στέλνουμε τέτοιο μήνυμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα. Αν υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι φταίνε, θα πρέπει να υποστούν τι κυρώσει. Εκεί πρέπει να είμαστε μετακίνητοι. Αυτά. Ανοίγουμε τη συζήτηση. Εγώ υπερασπίζομαι με την παρουσία μου εδώ ολόκληρο το ψήφισμα και όχι μόνο το ένα κομμάτι ενώ το άλλο το απορρίπτω, διότι δεν θέλουμε να λειτουργούμε έτσι. Μιλώντας δημοκρατικά, να σας υπενθυμίσω το ψήφισμα αυτό. Ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, με εξαίρεση 10 ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι δική τους ευθύνη. Αλλά η ευθύνη τώρα των υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να καταστήσουν σεβαστά τα κείμενα, τα πολιτικά κείμενα που ψήφισαν, που υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτέ. Δεν μπορεί να λέει η διοίκηση το, αυτό το κομμάτι το δέχομαι και αυτό όχι. Αν δεν πράξουν έτσι, πραγματικά σα υπόσχομαι, εγώ ίδιο θα παρέμβω is or not Οπότε, α, μας καθησυχάζει ή όχι το ότι ο δημόσιος τομέας αντικατοπτρίζει την ε, κοινωνία την ευρύτερη. Αλλά υπάρχει αυτή η ευθύνη που επομίζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι να αποτελέσουν παράδειγμα για την κοινωνία που θέλουμε. Λοιπόν, όλοι θα μιλήσουν, αλλά θα πάμε με τη σειρά. Κατόπιν, λοιπόν, έχουμε την Ίνγκε Μπέλ από την Γη των Γυναικών ε, στην Γερμανία. Πείτε μας για την οργάνωσή σας και πώς ιδρύθηκε. Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα είμαι εδώ πέρα με δίτο ρόλο. Πρώτα απ' όλα ως αντιπρόεδρο της οργάνωσης ε, Femme, η μεγαλύτερη οργάνωση δικαιωμάτων των γυναικών στην Γερμανία με γαλλικό όνομα όταν είχε ιδρυθεί τη δεκαετία του 80 από μια ομάδα γυναικών το όνομα το βρήκαν από το Τερντεζόμ βεβαίω, τη γη των ανθρώπων και κατά αναλογία έγινε το Τερντεφάμ είναι όμως μια γερμανική οργάνωση παρόλα αυτά η μεγαλύτερη στην Γερμανία Έχουμε γύρω στα 2.500 μέλη και άλλους τόσους υποστηρικτές ε, και γύρω στις 40 ομάδες ανά την Γερμανία σε πόλεις, ε, σε πανεπιστήμια όπου συγκεντρώνονται οι γυναίκες και κάνουν ε, κάποιες καμπάνιες εκστρατείας, αυτό κάνουμε βασικά. Είμαστε μια ΜΚΟ η οποία στηρίζει τα κορίτσια και τις γυναίκες ε, και τα δικαιώματά τους μέσω εκστρατιών, ενημέρωσης, ε, διεθνούς δικτύωσης ε, και προσωπικής βοήθειας και επίσης κάποια έργα αυτοβοήθειας στο εξωτερικό και εστιάζουμε σε πέντε τομείς τον γενετήσιο ακροτηριασμό Έχουμε στη Γερμανία 58.000 γυναίκες που επηρεάζονται από το θέμα αυτό, που έχουν υποστεί δηλαδή, ακροτηριασμό. Και υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή 13.000 κορίτσια κινδυνεύουν να υποστούν ακροτηριασμό ε, που ζουν στη Γερμανία και κινδυνεύουν να υποστούν ακροτηριασμό στις χώρες της τους. Έχουμε αυτό λοιπόν, έχουμε τους καταναγκαστικούς γάμους, την οικογενειακή βία και βεβαίως την σωματεμπορία και την πορνεία. Και όταν ακούμε στις ε, Βρυξέλλες, ε, όταν έρχομαι εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ε, θυμάμαι την εποχή που ήμουν δημοσιογράφος. Θα σας πω μετά γι' αυτό. Όταν είχα συναντήσει μια κοπέλα από την Βουλγαρία, ένα κορίτσι ανήλικο, που εκδιδόταν εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο γιατί ακολουθούσε τους ε, βουλευτές και μου έλεγε ανατριχιαστικές ε, λεπτομέρειες με το τι συνέβαινε γιατί δεν ε, την ήθελαν το βράδυ οι βουλευτές αλλά πριν ξεκινήσει η δουλειά το πρωί. Ενδιαφέρον λοιπόν είναι για σας να κάνετε και μια έρευνα για το τοπίο της ε, πορνείας ε, γύρω από το, τα θεσμικά όργανα εδώ και στις Βρυξέλλες γιατί ε, υπάρχουν πολλές γυναίκες που έχουν εξαναγκαστεί να εκδίδονται. Λοιπόν, κλείνω τα 50 σήμερα. Όχι, όχι σήμερα, όχι σήμερα, εντάξει ενώ ότι έχω περάσει τα 50. Στο πρώτο μισό της ε, ζωής μου ήμουν δημοσιογράφος στο πρώτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης ε, της Γερμανίας, ε, το ARD. Είχα γεννηθεί στην Ρουμανία, η μάνα μου με πήρε μαζί της και κατέφυγε στην Γερμανία όταν ήμουν τεσσάρων, αλλά βεβαίως τα Βαλκάνια ήταν πάντα μέσα μου και όταν έπεσε το τείχος ειδικεύτηκα σε σλαβικές γλώσσες και την ε, ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης ε, και ασχολήθηκα ως ανταποκρίτρια για τις χώρες των Βαλκανίων. Μίλα βουλγαρικά και ρουμανικά και βεβαίως έκανα ρεπορτάζ για αυτές τις χώρες. Και εκεί κάπου μέσα και τέλος δεκαετίας 90 και μέχρι το 2000 και επανέρχομαι στο 2000 ε, όχι για να σας λέω παλιές ιστορίες απλά να σου πω κάτι το οποίο με επηρεάζει και σήμερα. Ε, ήταν ε, η εποχή του πολέμου του Κοσμοπεδίου, μόλις είχε τελειώσει και οι βομβαρδισμοί μόλις είχαν ε, τελειώσει και είχα βρεθεί εκεί ως πολεμική ανταποκριτής. Επί τη ευκαιρία ποιος από εσά επίσης έχει πάει σε πολέμους και εργαστεί ως πολεμική ανταποκριτής. Καμία, κανείς. Μία Μία, δύο. Κάνα άντρα, όχι. Ε, και μία στο προηγούμενο πάνελ, μία κύρια. Όπως ξέρετε, πολεμική ανταποκριτής ε, ε, είναι σπάνιο πράγμα, πρόκειται για ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα. Εγώ ήμουν μία από αυτές που είχα πάει στον πόλεμο του Είχα σοκαριστεί πραγματικά ε, και πραγματικά δεν τα έχω ξεχάσει, με έχουν επηρεάσει μέχρι και σήμερα αυτά τα οποία είδα, η σωματεμπορία και η σεξουαλική εκμετάλλευση από τους στρατιώτες μετά τους βομβαρδισμούς, αφού τελείωσε ο πόλεμος, ήρθαν πολλοί στρατιώτες του ΟΗΕ, χιλιάδες, ε, σε κοσμοπέδιο και γουδμού για ως ειρηνευτικά στρατεύματα με τα γνωστά, τη γνωστή αποστολή. Και τι έκαναν. Πήγαιναν σε εκατοντάδες ανήλικα κορίτσια που είχαν εξωθηθεί στην ε, πορνεία, που είχαν έρθει από ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, Λευκορωσία, Ουκρανία, Βουλγαρία κτλ. Για να ε, τις εκμεταλλευτούν εκεί σεξουαλικά οι Και οι Γερμανοί στρατιώτες επίσης ε, χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες τους. Ε, και οι συνάδελφοί μου, οι άντρες, ε, δεν τα έλεγαν αυτά. Και είχα βρει εγώ ένα κοριτσάκι 14 ετών από τη Βουλγαρία που ήταν ένα από τα θύματα σε έναν οίκο ανοχής, παγιδευμένη εκεί και εκεί πέρα πήγαιναν οι Γερμανοί στρατιώτες της δύναμης, της Κέιφορ και έκανα ένα ρεπορτάζ. Δεν μπορούσα να το πιστέψω και δεν μπορούσα να πιστέψω γιατί δεν το έβλεπε κανείς, γιατί δεν το λέει κανείς άλλος. Ε, η απάντηση ήταν προφανής γιατί εντάξει ήταν ε, ανδρική υπόθεση το να είσαι πολεμική ανταποκριτή, αλλά ήταν και οι συνάδελφοί μου πελάτες. Ε, έκανα το ρεπορτάζ και όπως ξέρετε από τα ΜΜΕ ήταν μεγάλη αποκάλυψη, έγκλημα, σεξ, πόρνε, στρατιώτε, γερμανοί στρατιώτε. Έγινε λοιπόν σκάνδαλο εκεί πέρα το 2000 και τι είπε το Υπουργείο Άμυνας. Είπαν ε, όχι, οι Γερμανοί στρατιώτες δεν κάνουν τέτοια πράγματα και δεν ε, πάνε σε οίκους ανοχής, ε, πολύ περισσότερο με ανήλικα κορίτσια. Τους αρκεί το όπλο. Και σιγά σιγά λοιπόν πέρασα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, είχα κάνει τις ε, επαφές μου, όλοι ξέρουμε ότι έχουμε επαφή με πολιτικούς, δικαστές, ε, επιχειρηματίε κτλ. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω διάφορα ανθρωπιστικά έργα για τα κορίτσια αυτά που ήταν θύματα της σωματεμπορίας και να μπορέσουν να βρουν κάποια ζωή μετά και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Τελικά λοιπόν έφυγα από τη δημοσιογραφία, μπήκα περισσότερο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα είμαι στην άλλη όχθη, στην άλλη πλευρά με την οργάνωση αυτή, Third και δίνω συνεντεύξεις. Και τι συμβαίνει τώρα, το 2018 έχουμε το σκάνδαλο Oxfam. Ε, ανθρωπιστική οργάνωση υποτίθεται, αλλά όχι μόνο η Oxfam ε, και οι γιατροί χωρίς σύνορα ε, και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η ΚΕΡ, η UNICEF, όλοι αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί έχουν τα σεξουαλικά τους σκάνδαλα. Το προσωπικό τους κάνει ε, πάρτι και όργια με ιερόδουλες, ε, ανήλικα, παιδιά, σε περιοχές που πλήττονται από καταστροφές και πόλεμο, όπως στην Αϊτή. Αυτό ίσχυε ήδη το 2000 όταν ήμουν εγώ στο Κοσμοπέδιο, γιατί δεν ήταν μόνο οι στρατιώτες του ΟΗΕ που πραγματικά είχαν απογειώσει τους ε, οίκους ανοχής και τα λοιπά, σε Κοσμοπέδιο, Πουγουδουμού και σε αυτές τις χώρες που θεωρητικά απαγορεύεται η πορνεία. Αλλά βεβαίω κανεί δεν έκανε τίποτα. Οπότε δεν ήταν μόνο οι στρατιώτε του ΙΕ. Ήταν και οι ανθρωπιστικέ οργανώσει, η ΜΚΟ. Πήγαιναν εκεί πέρα, πλήρωναν για τις ας πούμε υπηρεσίες αυτές των ανήλικων ε, παιδιών και τότε υπήρχε αυτή η συλλογική σιωπή. Κανείς δεν το έλεγε, μόνο εγώ το είπα και τελικά ο ΟΗΕ εισήγαγε μια πολιτική μηδενικής άνοχης ε, όταν είναι στο εξωτερικό για ειρηνευτικές αποστολές ε, και έχουν και έναν κατάλογο απαγορευμένων ε, επιχειρήσεων, μπαρ, nightclub κτλ. που απαγορεύεται να πάνε ε, το προσωπικό του ΙΕ. Καμιά φορά όμως το προσωπικό βλέπει τον κατάλογο και θεωρεί ότι είναι να τα καλά τα μέρη, εκεί θα πάμε. Γιατί σας τα λέω αυτά. Το καιρό εκείνο, πριν από 18 χρόνια, κανείς δεν το έλεγε, ήταν ένα ανοιχτό μυστικό, όσοι ήταν εκεί το έβλεπαν και ήξεραν ότι και τα ειρηνευτικά στρατεύματα και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, ε, οι άντρες ε, πήγαιναν ε, εκεί πέρα, κατέφευγαν πορνεία. Τώρα 18 χρόνια μετά δεν είναι πια μυστικό, έχει βγει στο φως, οπότε μιλάμε γι' αυτό. Οι καιροί άλλαξαν και ήγκηκαν η ώρα. Έχει τελειώσει η ώρα Τη σεξουαλική ε, παρενόχλησης και σήμερα πλέον δεν θα έλεγε κανένα Υπουργείο όχι οι Γερμανοί στρατιώτε δεν πηγαίνουν στα πορνεία. Υπάρχουν τα σκάνδαλα, κάνουν τις εκστρατείες ενημέρωσης ε, και κάθε ένα από αυτού του οργανισμούς έχει κώδικα συμπεριφοράς και το προσωπικό του είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί τον κώδικα συμπεριφορά. Αλλά ξέρετε, όταν είναι εκεί πέρα μακριά από το σπίτι τους ε, και είσαι ο άντρας, ο λευκός, με λεφτά, με εξουσία, δεν σε βλέπει κανείς, ε, κανείς δεν θα καταλάβει στη χώρα σου τι γίνεται. Α, πας λοιπόν, σπάς τους κανόνες και έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή να τελειώσουμε αυτό το θέμα και ακριβώς ε, σε εσά επαφίεται ε, στις πρώην συναδέλφους μου και πραγματικά μου αρέσει η μαγεία αυτού του επαγγέλματος. Είναι τόσο ωραία δουλειά. Γιατί σε εσά επαφείτε λοιπόν τις γυναίκες να μην κάνετε τα στραβά μάτια, να δείτε, να ακούσετε και να δράσετε. Να κάνετε οι ερωτήσεις και μετά να δράσετε με αυτά τα οποία έχετε. Εσείς που είστε στα μήμη έχετε τόσα πολλά πράγματα, τόσα εργαλεία στη διάθεσή σας. Έχετε το ακροατήριο που είναι δικό σας. τα δικαιώματα των γυναικών ε, δεν ε, θεωρούνται δεδομένα. Πολύ εύκολα αφαιρούνται. Υπάρχει το δεξιό λαϊκιστικό κίνημα και το φεμινισμό έτσι, δεν τους ε, έρχεται και πολύ φυσικά. Δείτε λοιπόν αυτά τα ζητήματα, αντιμετωπίστε τα, δείτε το θέμα της πορνείας, της οικογενειακής βίας, τον ανισότητα των δύο φύλων, την ανισότητα στις αμοιβέ. Αυτό είναι ακριβώς ε, ο λόγος ε, για την ανισοκατανομή της ισχύω που βλέπουμε μεταξύ ανδρών και γυναικών. Λοιπόν, κοιτάξτε, ακούστε, ρωτήστε και δράστε. Ευχαριστώ. It's been a... Υπέροχα. Είμαστε εδώ δημοσιογράφοι. Είναι κάτι που θα έχω στο μυαλό μου για πάρα πολύ καιρό. Τις αλλαγές Υπήρχε οικονομική κρίση στις ε, Βρυξέλλες και άλλαξαν πολλά πράγματα με αυτήν. Αλλά αυτά που είπες ακριβώς μου θύμισαν εκείνον τον καταγγέλτη για αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Το θέμα μας σήμερα είναι δύναμη στις γυναίκες. Και το μήνυμα που ακούσαμε από εδώ ήταν ότι δύναμη έχουμε. Το θέμα είναι πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη. Υπάρχει εδώ μια νέα γυναίκα που την έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη για πάρα πολλά πράγματα. Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας σήμερα, να μας πείτε Συγγνώμη, συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι προηγουμένως. Ε, θα ακούσουμε ερωτήσεις μετά. Μα έχει να κάνει με τα προηγούμενα. Όταν θα έχει ολοκληρώσει το πάνελ της εισηγήσεις του, λέει συντονίστρια, τότε θα περάσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Σέριλ. Θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για την εμπειρία μου στην Ολλανδία όσον αφορά το φεμινισμό και τη δύναμη στα χέρια των γυναικών. Έχω κάποιες σημειώσεις. Εγώ θα σας μιλήσω για τη δομή της εξουσίας. Και αυτή των γυναικών είναι μία. Έχουμε φωνή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χώρο που έχουμε στη διάθεσή μας μέσα στην κοινωνία αλλά η κοινωνία πρέπει να λάβει υπόψη της αυτά που εμείς λέμε. Λοιπόν, είμαι η Χάτζη Αρμπενιλότη, είμαι 28 ετών από το Άμστερνταμ. Ήμουν δημοσιογράφος για 12 χρόνια, σε αρθρογραφούσα δηλαδή, σε εφημερίδα. Και για να φτάσω εκεί βέβαια χτύπησα πολλές πόρτες και τελικά ε, βρήκα δουλειά σε μεγάλες ε, εφημερίδες Οπότε εκεί ύψωνα τη φωνή μου, αλλά 12 χρόνια δούλεψα εκεί, τηλεόραση όμως, ραδιόφωνο, πουθενά δεν βρήκα χώρο που να δημοσιεύει τα πράγματα τα οποία εμένα με ενδιαφέραν. Αυτό ήταν βέβαια δικιά μου εμπειρία, αλλά όχι μόνο η δικιά μου, γιατί και γύρω μου άλλοι δημοσιογράφοι τελικά αναγκαζόντουσαν να γράψουν άρθρα τα οποία δεν ήταν ακριβώς αυτά τα οποία τους ενδιέφεραν. Τι είναι αυτό που είναι για μας, δεν είναι το Cosmopolitan, το Ascar, το CNN, τι είναι δηλαδή. Έπειτα, άρχισα να βλέπω ότι πολλοί λέγανε «Α, αυτά που γράφεις είναι φεμινιστικά». Λες και ήταν μια κακιά λέξη. Εγώ το βλέπω βέβαια σαν κομπλιμέντο, οπότε άρχισα να σκέφτομαι Μήπω τελικά πρέπει μαζί να αποφασίσουμε για το τι είναι ο φεμινισμό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει 2011 και ήταν 12 και να μην έχουμε συμφωνήσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο πρότυπο για τον φεμινισμό και για τις νέες γυναίκες. Οπότε με 10 χρόνια εμπειρία, σχέσεις και μεγάλο στόμα σκέφτηκα τότε ε, θα μπορούσα πια να μάθω, θα διαβάσω βιβλία για startups, θα μιλήσω με επενδυτές και θα ξεκινήσω μια πλατφόρμα. Δεν ήταν τόσο εύκολο, μου πήρε τρία χρόνια η όλη διαδικασία. Και μπήκα σε τόσα διοικητικά συμβούλια, ε, να ακούσω τόσους άντρες που μου λέγανε «Μπα, η δικιά σας ιδέα δεν είναι τόσο για σήμερα». Δεν σταμάτησα. Προσπαθούσα να εξηγήσω και έβλεπα γύρω μου ότι υπήρχαν και γυναίκες πολλές γύρω μου που θέλουν να πούν τα ίδια πράγματα με μένα. Οπότε είπα, γιατί να μην απευθυνθώ σε αυτές τις γυναίκες καλύτερα, ακόμα και αν στην αρχή δεν θα βγάζουμε λεφτά, μπορούμε όμως μαζί να οργανώσουμε ένα κίνημα, να σιγά σιγά έτσι να μπούμε και στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ακροατήριο θα έχουμε. Δεν μπορεί και έφτιαξα αυτήν την πλατφόρμα vilena.com. Ξεκινήσαμε καμιά κατοστή, ίσως λίγη παραπάνω. Πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε, είχαμε 600 που μας παρακολουθούσαν ήδη από την αρχή, χωρίς διαφημίσεις. Αυτό μας έδωσε πολύ θάρρος. Πολλοί περίμεναν κάποιου τέτοιου είδους πλατφόρμα. Και τι εννοώ τέτοιου είδου. Εννοώ μια μεγάλη ομάδα έξυπνων γυναικών που ξέρουν να γράφουν και που δημοσιεύουν κάτι κάθε μέρα. Σήμερα ο φαμινισμός δεν έχει να κάνει μόνο με τη σεξουαλική παρενόχληση ή μόνο με πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Όχι. Πρόκειται για μια δομή που έχουμε σε ολόκληρο τον κόσμο και που καθορίζει κάθε πτυχή της κοινωνίας μας. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα, αλλά σημαίνει επίσης ότι υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία δεν τα έχουμε ψάξει αρκετά. Δεν τα έχουμε χτενίσει αρκετά. Είχαμε πολλές περίπλοκες ε, συζητήσεις για πολλά θέματα και κατέληξαμε στο ότι έπρεπε να δημοσιεύουμε κάτι κάθε μέρα. Ε, συμπυκνωμένο, ε, με τρόπο που να ασχοληθούν και τα μεγάλα μέσα Μετά τον πρώτο χρόνο είχαμε 20 ε, δημοσιογράφους που μπόρεσαν από δικιά μας την πλατφόρμα να πάνε και στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Ήταν πάρα πολύ θετικό αυτό. Γίναμε και η μεγαλύτερη φεμινιστική πλατφόρμα στο Benelux. Η εμβέλειά μας ήταν ε, μεγαλύτερη, αλλά και το περιεχόμενό μας. Αυτά τα δύο χρόνια, λοιπόν, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, 7 μέρες τη βδομάδα, οργανωθήκαμε χωρίς να πληρωνόμαστε για να αντιγωνιστούμε, για να ανεβάσουμε τον πύχη όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης. Και είναι απογοητευτικό βέβαια να βλέπει κανείς ότι τελικά τα μέσα ενημέρωσης αντιγράφανε τα δικά μας θέματα, και ό,τι θέλανε χρησιμοποιούσαν, βγάζανε λεφτά από αυτά και συνεχίζανε με τον παραδοσιακό τρόπο για μένα στις κάτω χώρες, γράφω άρθρα γνώμης και άμα θέλω να βρω δουλειά, έτσι, μόνο 15-16% γράφουν τέτοια άρθρα και είναι βέβαια λευκές, έτσι. Αν ψάξουμε για έγχρωμες δεν θα βρούμε τίποτα περίπου. Και ακριβώς αυτό είναι που θέλω να υπογραμμίσω εδώ. Σήμερα Κοιτάξτε, συγκινήθηκα νωρίτερα σήμερα το πρωί όταν είδα τις νέες ε, ε τις Είπα πόσα πράγματα έχουν αλλάξει αυτά τα δύο χρόνια. Πριν από δύο χρόνια, εντάξει, υπήρχαν φυσικά φεμινιστές. Μετά τον Τραμπ όμως, το Me Too, ε, όταν ε, ξέρουμε ποια ήταν λέξη της χρονιάς και τα λοιπά, τελικά βλέπουμε ότι οι γυναίκες καταφέρνουμε να δούμε μία την άλλη και να αποφασίσουμε μαζί για το τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε μέσα από τους ανθρώπους εξουσίας για να μας συγκρίνουν. Όπως είπε και ο κύριος Μαρτέα νωρίτερα, εξακολουθούν οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία να παίρνουν τις αποφάσεις. Τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι σημαντικό. Και πράγματι τα περισσότερα έχουν να κάνουν με το πόσο αποδοτικό είναι κάτι οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι τελικά το φεμινισμό μας δεν πρόκειται να το εγκρίνει καμία εξουσία εφόσον είναι ανδροκρατούμενη. Εμείς οι ίδιες πρέπει να το κάνουμε. Και όπως λέμε συνήθως, ο δικός μας ο φεμινισμός πρέπει να είναι και στα δύο φύλλα ή αλλιώς δεν θα προχωρήσει. Όπως κάναμε για το ρατσισμό, όπως κάνουμε για τις διακρίσεις σε βάρος ηλικιωμένων. Θα μπορούσαμε να είμαστε εξαιρετικοί ηγέτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως για την πλατφόρμα μας, αφού δημοσίευσαμε 950 άρθρα, τα τρία προβλήματα τα οποία προέκυψαν για τις γυναίκες σήμερα, όπως το βλέπουμε εμείς, είναι πρώτον ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με το σώμα των γυναικών, δηλαδή σεξουαλική βία, δεν παίρνεται πάντα στα σοβαρά, και ο ιατρικός κόσμος είναι προσανατολισμένος ανδροκρατούμενος. Ό,τι έρευνες γίνονται ε, στρέφονται στους άντρες. Εμάς δηλαδή μας έχουν σαν ε, δεύτερης κατηγορίας ε, ασθενείς. Το δεύτερο πρόβλημα για το οποίο έχουμε γράψει πολύ είναι η οικονομική ισότητα. Δεν μπορεί βέβαια να πεις απλώς Όπω λέγαμε για καιρό, οι γυναίκε πρέπει να δουλεύουν σκληρά, να πιστεύουν στον εαυτό τους, έχουν δύναμη, θα τα καταφέρουν. Όχι, γιατί εδώ δεν πρόκειται για μια ατομική διαδικασία. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνει κάθε μια μας ατομικά και κατά πόσο θα καταφέρει να την ε, λάβουν σοβαρά η υπόψη η συναδελφή της ή όχι. Όχι. Το θέμα είναι πώς θα προβληθεί, γιατί τα πρότυπα είναι αντρικά. Γίνεται λοιπόν έρευνα και αυτή την έρευνα που γίνεται πρέπει να την πάρουμε σοβαρά. Ποιοι είναι οι κοινολογικοί παράγοντες. Έχουμε τρεις μέρες ε, πατρική άδεια στην Ολλανδία, ας πούμε. Δεν βοηθάμε τις γυναίκες να είναι οικονομικά ισότιμες. Ουσιαστικά Τις κατηγορούμε επειδή πρέπει να φροντίζουν το σπίτι και τα παιδιά τους. Για μας λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα να το δούμε και για τα δύο φύλλα το θέμα του φεμινισμού. Γίνονται περίπλοκες συζητήσεις, κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, αντίληψεις σε σχέση με το φεμινισμό Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένα προβλήματα και συγκεκριμένα θέματα. Στην πλατφόρμα μας θέλουμε να τα συνδυάσουμε αυτά. Δηλαδή, εντοπίζουμε το πρόβλημα, λέμε ποιος υποφέρει από αυτό το πρόβλημα, λέμε ποια θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά πάντα μιλάμε και για την ε, δύσκολη και περίπλοκη δομή που βρίσκεται πίσω από κάθε τέτοιο πρόβλημα και που είναι καλά δεδομένη στην κοινωνία μας. Και το τρίτο πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι το θέμα του ακτιβισμού και της δημοσιογραφίας, που πρέπει να επαναδιατυπωθεί. Οι δημοσιογράφοι ε, θεωρούν τους αυτούς ως αντικειμενικούς. Όμως, με τόσους άντρες στη δημοσιογραφία, δεν μπορεί να είναι αντικειμενική η εικόνα που δίνεται. Και έπειτα υπάρχει αντικειμενικότητα. Και μόνο που διαλέγει κανείς ένα θέμα για να δημοσιογραφήσει πάνω σε αυτό, κάνει μια επιλογή. Για να είναι τα μέσα ενημέρωσης πιο αντικειμονικά, πρέπει να είναι και πιο ε, ποικιλόμορφα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τους αναγνώστες μας. Δεν είμαστε απόλυτα αντικειμενικοί. Διαλέγουμε ένα θέμα, είναι επιλογή μας αυτή. Η δημοσιογραφία λοιπόν ε, μπορεί να κερδίσει από τον ακτιβισμό γιατί οι ακτιβιστές είναι ειδικοί, οργανώνονται αποτελεσματικά, φροντίζουν η αλλαγή να γίνει για αυτό που θέλουν και συγχρόνως οι ακτιβιστές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο άπαξ και τους δοθεί ευκαιρία να μιλήσουν πιο ανοιχτά με τους δημοσιογράφους. Φυσικά και θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν τη δημοσιογραφία, αλλά οι δημοσιογράφοι μπορούν να αποφασίσουν τι θα χρησιμοποιήσουν από αυτά. Αυτά είχα να πω, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Well, you said a lot. Είπατε πολλά και μας βρίσκεται όλους και όλες σύμφωνους. Να προσθέσω ένα-δυο πράγματα. Οι γυναίκες πράγματι, είμαστε βέβαια είναι καταπληκτικές, ε, καταπληκτικές ως ηγέτες και γι' αυτό το λόγο δεν μας αφήνουν γιατί είμαστε τρομακτικές. Οπότε μιλήσουμε γι' αυτό, το, για τον παράγοντο φόβο. Γιατί οι άντρες φοβούνται τις γυναίκες σε ηγετικές θέσεις. Γιατί είμαστε ακτιβίστριες είμαστε μαχητικέ ζητάμε να μάθουμε πράγματα, ρωτάμε δύσκολα πράγματα. Λέμε γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι. Αφήστε με να σας επενέσω λίγο σε αυτά που είπατε πρώτα. Διότι ε, ανοίξατε πολλά θέματα εδώ. Και κατά κάποιο τρόπο συνενώσατε τα διάφορα θέματα που συζητήσαμε σήμερα. Στον οργανισμό μας θα έχετε ακούσει για τα βασικά για τις βασικές ε, δεξιότητες, επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά. Και στην Αμερική λένε STEAM αντί για STEM, όπως λέμε στην Ευρώπη. Προσθέτουν δηλαδή και τις τέχνες και συνδυάζουν τον τομέα των καλών τεχνών με αυτές τις ισχυρές, τις δυνατές τεχνικές δυνατότητες και αυτό θα μας οδηγήσει στη μελλοντική μας οικονομία. και εγώ για το ε έλεγα entrepreneurship μπροστά την επιχειρηματικότητα και μιλάμε για e-steam το οποίο προωθούμε στις γυναίκες και στα κορίτσια και θέλω να σας συγχαρώ. Είστε ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνδυασμού τεχνολογίας, δημιουργικότητας, ενό σαφού μηνύματος, ένα σαφές όραμα αυτό που μας προτείνεται ως νέα γυναίκα για όλα αυτά τα πολύ δύσκολα θέματα αποτελείται ένα εξαιρετικό μοντέλο για τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους του κόσμου αυτού. Συγχαρητήρια λοιπόν για σας. Ωραία. Ωραία, ας ε, στεγνώσω τα δάκρυά μου και ξέρω ότι μας περιμένουν πολλές ερωτήσεις ε, από το κοινό. Παρακαλώ, από πίσω. Είναι εδώ ακόμη η κυρία που ήθελε να κάνει την ερώτηση. Λέγομαι Λίλια Ηλίου, είμαι από τη Βουλγαρία από το περιοδικό ΕΒΑ. Πήγα και είδα κατά πόσο είναι νόμιμη πορνεία στη Βουλγαρία. Δεν είναι. Και αυτό είναι σημαντικό αυτό που είπαμε. Ενώ είπατε το αντίθετο πριν. Είναι σημαντικό να υποθεί λοιπόν αυτό. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είπατε ότι η πορνεία είναι νόμιμη. Είπε κάποιο, αλλά δεν είναι. Όχι εγώ είπα ότι δεν είναι νόμιμη. Α, ζητά συγγνώμη κύριε Αποτοκίνο, Δεν κατάλαβα σωστά. Είναι παράνομη λοιπόν η πορνεία στη Βουλγαρία. Ωραία. Ούτε εκεί είναι νόμιμη, ούτε στην Ρουμανία, ούτε στο Κοσφοπέδιο, ούτε στην Πογοδομού, ούτε πουθενά. Η διπλανή σα κυρία έχει μια ερώτηση. Εγώ έχω ένα σχόλιο ουσιαστικά. Ήθελα να μιλήσω για τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, αλλά πριν από αυτό, εμπνευσμένη από τα όσα είπατε για του βιασμού, ήθελα να σα πω ότι Ξέρετε, οι βιασμοί στον πόλεμο ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα και στο Κωσυφοπαίδιο και στην Κροατία από όπου προέρχομαι εγώ. Εργάζομαι για ένα πολιτικό περιοδικό, το National. Και ξέρετε, χρειάστηκαν 20 χρόνια για τις γυναίκες που βιάστηκαν στον τελευταίο πόλεμο ώστε να αρχίσουν να το συζητούν. Και λόγω του βιβλίου όπου δημοσιεύτηκαν οι ιστορίες τους, εκείνη την εποχή εγώ εργαζόμουν για τον πρόεδρο της ε, Κροατίας Σοσιαλδημοκράτη και τότε ήταν η πρώτη φορά που τους δόθηκε ο χαρακτηρισμός ε, ε, άμαχων θυματών του πολέμου. Και εκεί πήγαμε στον Ποκοβαρό που βιάστηκαν οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες και προωθήθηκε ένα νομοθέτημα βάσει του οποίου η Δημοκρατία της Κροατίας τώρα πρέπει να ε, πληρώσει για την ε, ψυχολογική και σωματική τους αποκατάσταση και λαμβάνουν κάποιο ε, ποσό ως βοήθεια από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ανακοινώσω, αφού μιλάμε για φεμινισμό, αύριο είναι η Διεθνή ημέρα των γυναικών και πολλές φεμινιστικές μικιό στην Κροατία σε τρεις πόλεις θα δράσουν με σκοπό να ασκήσουν πίεση στην κρατική κυβέρνηση για να κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και παρότι ο Πρωθυπουργό έχει αρκετή δύναμη στο Κοινοβούλιο για να το πράξει, διστάζει. Γιατί, διότι η αντίσταση έρχεται από, όχι από τους δικούς του τους ακροδεξιούς, αλλά από άλλες ομάδες πιο προοδευτικές υποτίθεται και το δικό του κόμμα ανήκει στο ΕΛΚ και παρότι ξέρω ότι το ΕΛΚ ψήφισε υπέρ του ψηφίσματο για την κύρωση του τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη πέρσι, τα περισσότερα μέλη του ΕΛΚ δεν το έπραξαν. Τι παρατηρούμε λοιπόν, μια κατάσταση παρόμοια με αυτή στην Πολωνία. Στην Κροατία κλήθηκαν όλοι ε, διάφοροι ε, υποστηρικτές, ε, υποστηρικτές τους να μην ψηφίσουν και αυτοί φυσικά επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Παρότι λοιπόν δεν είναι υποχρεωτικό, το 96% των παιδιών πηγαίνουν ε, σε αυτά τα θρησκευτικά μαθήματα. Πηγαίνουν στο κατηχητικό και τι τους μαθαίνουν εκεί για τις γυναίκες ότι πρέπει να τηρούν ε, τον παραδοσιακό τους ρόλο, το να γίνουν μανάδες κτλ και εκεί τους ειδοποιούν τα παιδιά για τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη, γιατί αναφέρουν ότι παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το φύλλο. Αυτό του ενοχλεί, το φύλλο και το σεξ και φοβούνται ότι αυτή η σύμβαση θα χρησιμοποιηθεί για δεν ξέρω ποιους σκοπού. Συγγνώμη που μακρηγορώ, απλά ήθελα να πω κάτι για τη βία, για την ενδοοικογενειακή βία Παρότι η κρατική νομοθεσία είναι επαρκής και παρέχει αρκετά εργαλεία στο δικαστικό, εφόσον θελήσει να την υλοποιήσει, παρόλα αυτά παρατηρείται αύξηση της βίας. Περίπου 300 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους ε, στα χέρια των ε, ανδρών συντρόφων τους ε, τα τελευταία χρόνια, 19 πέρυσι. Παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο με έναν υψηλό βαθμό πολιτικό σε τοπικό επίπεδο και πάλι μέλος του κυρίαρχου κόμματος του ΕΛΚ που η γυναίκα του τόλμησε να τον καταδώσει για ενδοοικογενειακή βία χρόνων και μάλιστα προσπάθησε να έρθει σε επαφή και με τον Πρωθυπουργό. Συγγνώμη να σας διακόψω γιατί είμαι βέβαιη. Ήθελα απλό να πω απλά ότι όταν τον κατέδωσε τελικά και άσκησε μήνυση αποφάσισε να αποσυρθεί, να αποσύρει γιατί την καταδίκασαν η γυναίκα της, η οικογένειά της, οι συγγενείς της, τα παιδιά της και το πολιτικό κόμμα άντρα της. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Τι είπατε. Θα απαντήσουν βέβαια εδώ οι διάφοροι συγκητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα υπουργό για θέματα ισότητας στην κυβέρνηση της Πολωνίας όταν ετοιμάσαμε τα διάφορα έγγραφα για την υπογραφή και την κύρωση τελικά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολη. Πάνω από δύο χρόνια τώρα έχουν περάσει από τότε που εμείς κυρώσαμε την συμφωνία αυτή. Δεν λέω ότι ήμασταν η πρώτη χώρα, αλλά ήμασταν μία από τι πρώτε ευρωπαϊκέ χώρε που το έκανε και η συζήτηση στην Πολωνία ήταν ίδια με αυτή που περιγράψατε. Η Εκκλησία ήταν κατά τη σύμβαση, γιατί ακριβώς αναφέρονταν ο όρος φίλο στην σύμβαση. Και ξεκίνησε μια ολόκληρη συζήτηση όσον αφορά το περιεχόμενο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα φύλλα και είναι μια συζήτηση που έγινε σε ε, πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ουσιαστικά δεν ήταν σαφές για πολύ κόσμο τι ακριβώς εννοούσαμε με τον όρο φύλλο. Και γι' αυτό σε πολλές χώρες δεν προχώρησε η σύμβαση αυτή, στη Βουλγαρία για παράδειγμα. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι στην αρχή ένα σημαντικό μέρος των πολιτικών και στη χώρα μου ήταν υπέρ της κύρωσης, μετά από τα διάφορα δημοψηφίσματα έγιναν στην Πολωνία σε διάφορους δήμους, διάφορες διασκέψεις, συναντήσεις με οργανώσεις και μετά τέλο πάντων από όλες αυτές τις συζητήσεις που κρατήσανε ώρες και ώρες και όπου ήταν παρόντες οι πιο σημαντικοί πολιτικοί, άλλαξε ο τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα και έτσι ετοιμάστηκε ένα πρώτο σχέδιο στο Κοινοβούλιο υπέρ της σύμβασης αυτής και μετά έγινε και η κύρωση. Θέλω να πω τα πράγματα δεν έγιναν εύκολα χρειάστηκε πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ προβληματισμό για να καταλήξουμε στην κύρωση αυτή που έγινε τελικά. Και κάτι ακόμα. Εγώ εκπροσωπώ το ΕΛΚ, μια χριστιανοδημοκρατική οικογένεια. Θέλω να σας πω ότι το ΕΛΚ είναι υπέρ της καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας και αγωνίζεται γι' αυτό. Ε, πρωτοστάτησαν οι βουλευτές μας σε εκθέσεις σχετικά με το θέμα αυτό όπου λέγαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσχωρήσει στη σύμβαση αυτή της Κωνσταντινούπολης. Είναι αλήθεια ότι δεν ήμασταν πολλοί. Δεν πρέπει λοιπόν να επιτίθεται κανείς. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Μαρτά τώρα για τις διαδικασίες στο Κοινοβούλιο. Η συνάδελφός μου, κυρία Μωρέ Σαρτιέ, είναι αυτή που ηγείται της ομάδας που εξετάζει τα θέματα παρενόχλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρότεινε οι ευρωβουλευτές κάθε φορά που έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αναλαμβάνουν δηλαδή, τα καθήκοντά τους εδώ, να υπογράφουν ένα κώδικα δεντολογίας. Τα θύματα όντως δεν πάνε ε, συχνά ε, σε αυτήν την ομάδα για να καταγγείλουν, γιατί όντως φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται και μια συζήτηση πιο άτυπη με την ομάδα αυτή. Αυτό που κάνουμε πάντω να ξέρετε ότι δεν έχει να κάνει με το κόμμα από το οποίο προερχόμαστε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και να πάψει να υπάρχει το φαινόμενο. Θα πω τώρα κάποια πράγματα και εγώ, όλες συντονίστρια, για τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη που έχει να κάνει με την απειλή τη βία. Και έτσι φτάνουμε και στο εικονικό περιβάλλον, τη ρητορική μίσους, στον κυβερνό χώρο, την ψυχολογική βία. Για να επανέλθουμε σε αυτά που ακούγαμε πριν. Ίσως εσείς θα θέλατε να αντιδράσετε, να απαντήσετε, κύριος Μαρτά, εσείς. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, Όντω δεν πρέπει να βλέπουμε αυτή τη διαφορά δεξιά-αριστερά. Είναι αλήθεια ότι ένα μεγάλο μέρο του ΕΛΚ συμφωνεί με αυτά που λέτε. Αλλά υπάρχει και ένα τμήμα του ΕΛΚ που δεν συμφωνεί με αυτή τη γραμμή και καλά κάνατε και το υπογραμμίσατε. Κάθε φορά που έχουμε ένα κείμενο για τα δικαιώματα τη γυναίκα και μιλάμε για τη σύμβαση του Κωνσταντινούπολη, λυπάμαι που το λέω, αλλά εσεί σαν δημοσιογράφοι μπορείτε να το περιτέψετε. Το ΕΛΚ βάζει μια κόκκινη γραμμή στο θέμα τη άμβλωση. Αν μιλάμε για το δικαίωμα στην άμβλωση, δεν το ψηφίζω. το, το ΕΛΚ όχι ένας ή ένα η τοποθέτηση και η θέση τη ομάδα. Οπότε ωραία, αυτά που λέτε εσεί ισχύουν, αλλά δεν ήσασταν η πλειοψηφία στο ΕΛΚ. Και για το θέμα τη σεξουαλικής παρενόχληση εδώ, όντω η κυρία Σαρτιέ συμμετέχει στου κοσμήτορε και εκείνη δημιούργησε, όχι μόνη τη, βέβαια, αλλά είναι μία ε, από τους υπεύθυνου στην Επιτροπή αυτή που εξετάζει τα θέματα παρενόχληση, αλλά και εκείνη αντιδράει σε μερικά πράγματα για να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν λέω ότι είναι δικιά τη προσωπική θέση, έτσι, γιατί δεν το νομίζω αυτό, αλλά είναι θέση του ΕΛΚ που την εμποδίζει και που λέει, Α, όχι, δεν χρειαζόμαστε. Ο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριο Βέλε, για παράδειγμα, που είναι από το ΕΛΚ, είναι αυτό που λέει, Όχι, ποτέ δεν θα επιτρέψουμε εξωτερικό έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι γεγονό. Γεγονότα λέμε, δεν λέμε υποθέσεις. Ευχαριστώ κι εγώ. Θέλω να προσθέσω κι εγώ κάτι. Είναι ακριβώς το ίδιο το πρόβλημα. Επανέρχομαι σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα, την δομή της εξουσίας. Πρέπει να είμαστε μια κρίσιμη μάζα που θα φωνάξει, που θα πιέσει τις παραδοσιακές δομές εξουσίας. Θα κάνουμε πολλή φασαρία. Αν όμως παραμένουμε εκτός δομών εξουσίας, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Πραγματικά. Το έχω δει ξανά και ξανά οι γυναίκες να κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν αυτό τον αγώνα. Και κερδίζουν ατομικά, αλλά η πίεση που έρχεται απ' έξω είναι τόσο μεγάλη Το έχουμε αυτό το πρόβλημα στην πλατφόρμα μας, ε, το Βιλένο, ότι δηλαδή μιλάμε με πολιτικούς, οργανώνουμε εκδηλώσεις, χωρίς χρήματα, έτσι. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να σταματήσουμε να ξοδεύουμε τα χρήματά μας και το χρόνο μας για να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μας. Προτείνουμε λύσεις, αλλά θα πρέπει και οι παραδοσιακές δομές εξουσίας να μας προσφέρουν χώρο για τη συνεισφορά μας αυτή. Γιατί υπάρχει απόσταση ανάμεσα στους ανθρώπους και τους πολιτικούς, τα μέσα ενημέρωσης. Ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στη δημοσιογραφία, ούτε στους πολιτικούς. Υπάρχει ο ακτιβισμός που ξεκινάει, όπως με τα hashtag είδαμε, Πολλά μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σας πούμε που εντοπίσετε το πρόβλημα, να σα προτείνουμε λύσει Εμεί μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά για εσά αλλά αν ε, οι δομές εξουσίας δεν μας δώσουν χώρο για αυτά, δεν πρόκειται να καταλήξουμε πουθενά. Πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση σε πρωτοβουλίες. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν ήθελα εδώ να δημιουργήσω πόλεμο ανάμεσα σε δύο κόμματα, αλλά θέλω να πω ότι για μήνες ο άνθρωπος αυτός που σας είπα πριν ε, διακόπτει η συντονίστρια. Ναι, καταλάβαμε τι μας λέτε. Πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη. Το θέμα της αλληλεγγύης ε, των φίλων, σημαντικό, από το Οικονομικό Φόρουμ την προηγούμενη εβδομάδα έμαθα ότι οι ομάδες γυναικών είναι πιο διαφοροποιημένες από ότι ομάδες ανδρών. Και αυτό φαίνεται, το βλέπετε και εσείς στη δημοσιογραφία και στην πολιτική. Ακόμα και με διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις οι γυναίκες τα καταφέρνουμε μεταξύ μας να τα βρούμε και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε το φίλο μας. Συνήθως γίνεται, όχι πάντα βέβαια. Κάποια από τα εμπόδια στην ισότητα είναι βέβαια και γυναίκες, αν και είναι η εξαίρεση. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν και άντρες που μας βοηθάνε να πετύχουμε την ισότητα. Όπως είπε και ο κύριος Μαρτά, είναι προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας η ισότητα. Άλλη μια ερώτηση να ακούσουμε. Για τις 6 λεπτά έχουμε και το κλείσιμο, έτσι, η τελευταία εισήγηση. Και θα πρέπει να ακούσουμε και την ε, Ασιατζέντο. Ποιος έχει ερώτηση προς το πάνελ ή να προχωρήσουμε στο επόμενο. Βλέπετε, α, εσείς παρακαλώ, παρακαλώ κυρία Σόρτοβα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για την ισότητα ανδρών και γυναικών και μιλάμε επίσης και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα όμως δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Λυπάμαι που χωρίζουμε τα κόμματα δεξιά-αριστερά γιατί είναι θέμα συνείδησης και όλοι έχουμε μια συνείδηση. Πρέπει να τα σεβαστούμε τα δικαιώματα αυτά λοιπόν. Και το κοινό μεταξύ μας είναι η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η προστασία των γυναικών. Γι' αυτό και εγώ βρίσκομαι εδώ σε αυτό το σεμινάριο και γι' αυτό και ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές. Δεν ήταν ερώτηση, ήταν σχόλιο. Συντονίστρια, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά αυτή είναι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και νομίζω ότι μπορούμε να συνδέσουμε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των γυναικών με το μέλλον αυτού του μεγάλου πειράματος. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ και τα μέλη του πάνελ.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 ladies and ladies and gentlemen. May I please ask you to take your seats? Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Ε, συμφωνείτε όλοι μαζί μου ότι έχουμε μια τεράστια ευκαιρία στο τελευταίο κομμάτι της ε, πολύ ενδιαφέρουσας ε, ημερίδας μας σήμερα. Πώς σας φάνηκε μέχρι στιγμής? Ανταποκρίθηκε στις ε, προσδοκίες σας, ελπίζω ναι. Ίσως ανοίξαμε περισσότερα θέματα από όσα κλείσαμε, αλλά αυτό είναι δική σας δουλειά. Και πραγματικά είστε ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς κάνει κανείς τη δουλειά του. Αλληλεγγύη, στήριξη. Είναι δύσκολο να είναι κανείς κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είμαστε όλοι στο πλευρό σας. Ε, θα το διαπιστώσετε. Κυρίες και κύριοι, ε, θα παρουσιαστεί μόνη της, αλλά ε, να σας πω, πρόκειται για την Άζια Αρτζέντο. Thank you. Thank you. I wrote a story that's not... ευχαριστώ. Έγραψα μια ιστορία που δεν είναι για τους ε, λιπόψυχους ε, και ήταν δύσκολο να την γράψω. Και ζητώ συγγνώμη αν θα είναι δύσκολο να την ακούσετε, αλλά νομίζω ότι είναι αναγκαίο, ειδικά σήμερα. Άζια Αρτζέντο λέγομαι, σκηνοθέτης ε, και ηθοποιός, κόρη και μητέρα επιζών ε, σεξουαλικής επίθεσης ε, και ήρθα σήμερα να σας μιλήσω εκ βάθους καρδίας για την εμπειρία μου τον αντίκτυπο που είχε και το αποτέλεσμά της και για το κίνημα αυτό, το Me Too, στα κοινωνικά μέσα που έχει γίνει μια φοβερή δύναμη για τις γυναίκες παντού για να μιλήσουν, να πούν την αλήθεια, να ακουστούν, να τις πιστέψουν και το πώς με ενδυνάμωσε και εμένα με τρόπο που ποτέ ε, δεν φανταζόμουν. Ξεκίνησα ασθενή όταν ήμουν παιδί, από 9 ετών. Πάντα μου άρεσε ο κινηματογράφος, είναι η ζωή μου, η κληρονομιά μου, είναι στο αίμα μου, το πάθος μου. Όμως ε, συνειδητοποίησα από πολύ τρυφερή ηλικία ότι ο κινηματογράφος έχει μια αυστηρή ιεραρχία, μια πυραμίδα. Πάνω πάνω είναι η παραγωγή, μετά οι σκηνοθέτες και μετά οι ηθοποιοί και κάτω-κάτω οι γυναίκες. Ως ηθοποιός ε, και γυναίκα στον κινηματογράφο πριν ε, πάει κανείς ε, καν σε ένα στούντιο είναι σε θέση υποταγής σε σχέση με όλους τους άλλους άντρες. Παραγούς, σκηνοθέτες, άλλους τοπίους. Ακόμα και τους ατζέντιδες και τους δημοσιοσχεσίτες. Όλοι ασκούν πίεση πάνω σου με διαφορετικούς τρόπους πίεση για συγκεκριμένη συμπεριφορά, συγκεκριμένο ντύσιμο, για να πάρεις κάποιον ρόλο. Είχα καταλάβει ως παιδί ότι δεν είχα εξουσία εγώ στο γύρισμα, έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου, αυτό το οποίο μου λέγανε, δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανέναν και δεν μπορούσα να πω τίποτα σε κανέναν. Και βεβαίως ε, υπήρχε αυτή η θέση υποταγής που τελικά μεταφέρθηκε και στην πραγματική μου ζωή. Αν με αδικούσαν ε, σωματικά ή ψυχολογικά, δεν πίστευα ότι θα με άκουγαν ή θα με πίστευαν ή ότι είχε κάποιο νόημα να πω κάτι. Μεγάλωσα στα στούντιο, ενηλικιώθηκα στα στούντιο και όταν από παιδί έγινα έφηβος, μετά έγινα γυναίκα. Πάντα ήμουν δειλή, αλλά και αλητάκι. Έτσι, νομίζω τουλάχιστον. Αλλά επίσης ήμουν και άβολα στο σώμα μου, οπότε όταν έγινα έφηβος, ήταν ήταν δύσκολο για μένα να αποδεχτώ ότι ήμουν ε, ένα σεξουαλικό αντικείμενο. Δεν μου φαινόταν φυσικό. Και σιγά σιγά η ρόλη που μου προσφερόταν γινόταν πιο αισθησιακή, το ίδιο και οι χαρακτήρες που έπαιζα και συχνά απαιτήθηκε να εμφανίζομαι γυμνή. Και από αγοροκόριτσο έγινα σιγά σιγά, έπαιρνα ρόλους ε, σεξουαλικής ε, γυναίκας. Σιγά σιγά λοιπόν έγινα σεξουαλικό αντικείμενο. Μπορούσα να πω όχι. Είχα επιλογή. Ήξερα ότι δεν είχα επιλογή και αν ήθελα να δουλέψω έπρεπε να αποδεχτώ τους ρόλους που είχα διαλέξει για μένα. Και ήξερα πως οι γυναίκες στις ε, ταινίες είχαν δύο ρόλους. Είτε τη μητέρα είτε την πόρνη στην πραγματικότητα δεν υπήρχε επιλογή. Και ε, μετά οι ρόλοι που έπαιζα ε, επηρέασαν και την πραγματική μου ζωή. Ως μια νέα γυναίκα στην Ιταλία, όποτε πήγαινα σε μια φωτογράφηση για τις ε, ταινίε μου, υπήρχαν μόνο εσόρουχα και σεξι φορέματα. Πότε οι τουαλέτες που φανταζόμουν ότι θα φορούσα. Και έτσι στα μάτια του κοινού είχα μια δημόσια εικόνα ε, σεξουαλική. Όχι η μητέρα, η πόρνη. Αυτόν τον ρόλο μου έδωσαν να παίξω. Όταν ήμουν 20 ετών έκανα ακρόαση για μια ταινία ονόματι Be Monkey, η πρώτη μου ταινία στην αγγλική γλώσσα με έναν σκηνοθέτη που είχε πολλές υποψηφιότητε για Όσκαρ και όταν πήρα τον ρόλο πήγα και είδα τον πατέρα μου στο στούντιο και μου είπε «Άζια θα πάρεις Όσκαρ». Ήταν πολύ περήφανος για μένα. Και εγώ ήμουν περήφανη για τον εαυτό μου. Δεν ήξερα ότι τελικά αυτό θα μου τα στερούσε όλα. Τον Μάιο του 1997 πήγα στο φεστιβάλ των Κανών για την ταινία αυτή, όπου θα με εξέθεται η μοίραμαξη εταιρεία στα ΜΜΕ όλου του κόσμου. Και εκεί πέρα με βίασε 21 ετών ο Χάρβι Βάινσταϊν. Αυτός λέει ότι υπήρχε συνένεση. Ο δικηγόρος του λέει ότι ο Βάινσταϊν ε, δεν φταίει γιατί δεν εφήβρε αυτός ε, το casting ε, του καναπέ. Και επίσης, όπως είπε, αν μια γυναίκα κάνει σεξ για να προωθήσει την καριέρα της στο Hollywood, αυτό δεν είναι βιασμός. Ήρθα να σας πω σήμερα λοιπόν ότι δεν υπήρχε καμία συνένεση. Με γέλασαν, πήγα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο από έναν συνεργάτη του, μου είπαν ότι θα πήγαινα σε πάρτι, τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πάρτι για δύο, εμένα και τον εν λόγω. Και εκεί μέσα συνετρίβησαν όλα μου τα όνειρα. Νόμιζα ότι ήμουν σκληρή και έξυπνη, όμως είχα ηλίθιες ελπίδες. Ήμουν αμνός 21 ετών, νόμιζα ότι είμαι μια γυναίκα του κόσμου γιατί είχα πετύχει αρκετά πράγματα για την ηλικία μου, αλλά ήμουν απλά μια ηλίθια κοπέλα ως πρόβατο επισφαγή και το δέχτηκα αυτό ως ε, ρόλο μου, ως μέρος της δουλειάς μου. Αυτό νόμιζα ήταν, αυτό ήταν ο κόσμος ένας κόσμος σκληρός, ε, όπου και άλλες γυναίκες, τις οποίες θαύμαζα όλη μου τη ζωή, ε, και αυτές ήταν τελείως ανίσχυρες ε, στα χέρια των ανδρών. Αν μπορούσα να πάω πίσω σε αυτήν την νύχτα, δεν θα μπορούσα, δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτήν την πόρτα. Αυτό το οποίο συνέβη λοιπόν άλλαξε την ζωή μου για πάντα. Απογοητεύτηκα, με σημάδεψε απογοητεύτηκα από τη ζωή και τους ανθρώπους. Έκτοτε υποφέρω από κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες και συνειδητά και ασυνειδητά προσπάθησα να τιμωρήσω τον εαυτό μου, γνωρίζοντας ότι μόνο τον εαυτό μου έβλεπα. Όλη μου την ενήλικη ζωή είμαι σε ψυχοθεραπεία. Το τραυματικό αυτό γεγονός άφησε μια πληγή που ποτέ δεν έκλεισε ε, και δεν μπορούσα να μιλήσω για τον βιασμό μου ούτε με τους δικούς μου και τον ε, ψυχοθεραπευτή μου. Το είχα αποθήσει από τη μνήμη μου. Αυτή ήταν η άμυνά μου για να μην τρελαθώ. Και έλεγα ότι ποτέ δεν συνέβη και έβαζα το τέρας κάτω από το χαλί. Αλλά εκεί πέρα μεγάλωσε αυτό και έγινε τεράστιο. Έγινε ο ελέφαντας όπως λέμε στο δωμάτιο. Το θέμα για το οποίο δεν μιλάει κανείς. Απόθεσα λοιπόν αυτές τις μνήμες για να επιζήσω. Και βεβαίως, όπως μου λένε οι ψυχολόγοι, θα τις ανακτήσω. Αλλά έριχναν τη μακριά σκιά τους σε όλες μου τις σχέσεις, στη δουλειά, στην αγάπη, στο σεξ. Σταμάτησα να εμπιστεύομαι τον κόσμο. Πήγα και κλείστηκα στο καβούκι μου. Ε, φαινόμουν ακόμη πιο σκληρή, αλλά στην ουσία έλεγα ψέματα στον εαυτό μου, γιατί δεν ήθελα να αισθάνομαι ως θύμα. Είναι πολύ άσχημη η κατάσταση, αλλά χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια για να δεχτώ και να μπορέσω να πω σε κάποιον το τι μου είχε συμβεί. Και αυτό συνέβη λόγω του μύτου πριν ακόμα ε, γίνει γνωστό αυτό. Αυτό ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, 17 χρόνια μετά από την νύχτα στις ε, Κάνες. Ε, ήμουν 38 ετών, μητέρα δύο παιδιών πια μιλούσα σε μία φίλη που μου είπε τη δικιά της ιστορία, μια ιστορία τόσο παρόμοια με την δική μου που δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ταυτίστηκα με την εμπειρία της, ώστε για πρώτη φορά αισθάνθηκα την ικανότητα και την ανάγκη να της αποκαλύψω το προσωπικό μου τραύμα. Της είπα τα πάντα. Τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια. Και με άκουσε και με κατάλαβε. Και κλάψαμε και οι δυο μας. Μετά, τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, εντελώς ξαφνικά πήρε τηλέφωνο ένας δημοσιογράφος που δούλευε για το New Yorker, ο Ρόναλτ Φάιλερ. Δεν τον ήξερα. Έγραφε μια ιστορία για τον διαστημό τον άνθρωπο που με κακοποίησε και είχε ακούσει φήμες για μένα και είχε ανακαλύψει το μυστικό μου που ούτε οι κοντινοί μου φίλοι δεν ήξεραν και τότε συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά τα χρόνια εγώ κρατούσα την αλήθεια μυστικό πολλοί άνθρωποι ήδη γνώριζαν τι μου είχε συμβεί όχι μόνο ο αλλά και όλη η συνένοχή του ήταν μια αποκάλυψη που με σοκάρισε και με αναστάτωσε και με τρομοκράτησε. Συνειδητοποίησε ότι το είχαν συγκαλύψει και αποσιωπήσει, αλλά ήταν ένα ανοιχτό μυστικό που το λέγανε μεταξύ τους όλη την ώρα, μέχρι που τελικά έφτασε και στα αυτιά αυτού του δημοσιογράφου. Όταν αποφάσισα λοιπόν να μιλήσω για τον άνθρωπο που με κακοποίησε, να τον κατονομάσω και να μιλήσω επωνύμως στο New Yorker με την ιστορία μου, ήταν επειδή μου το επαγόρευσε η συνείδησή μου. Το πάλεψα. Σκέφτηκα την οικογένειά μου και πώς θα τους επηρέαζε για να αντιμετωπίσουμε. Το να αντιμετωπίσω αυτό το κακό ήταν ότι δυσκολότερο έκανα για να αντιμετωπίσω επίσης την ενοχή και την τροπή που ένιωθα τόσα χρόνια. Ήξερα ότι έπρεπε να ομολογήσω τα πάντα, τα ελαττώματά μου. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαμε να πείσουμε και τις άλλες γυναίκες ότι έπρεπε να μιλήσουν. Αυτός είναι ο φόβος που έχουμε πάντα ως γυναίκες. Ότι θα μας ασκήσουν κριτική, θα μας σπηλώσουν επειδή μιλάμε. Αυτό το φόβο είχα. Στην Ιταλία τις γυναίκες την δείχνει η τηλεόραση και τα ΜΜΕ μόνο ως σεξουαλικά αντικείμενα, όπως ήμουν και εγώ όλη μου την ενήλικη ζωή. Και όταν πουν αυτά τα οποία σκέφτονται, δαιμονοποιούνται. Είναι σεξιστική εντελώς η Ιταλία και θεωρεί ότι ο μισογυνισμός είναι κάτι το φυσιολογικό και όταν σκοτώνει, ένας, σκοτώνει κάθε τρεις μέρες ένας ε, άντρας ε, μία γυναίκα και πολλές γυναίκες φύστανται σεξουαλική βία. Μέχρι το 1981 οι κατηγορίες του βιασμού απορρίπτονταν εάν ε, ακολουθούσε γάμος ο λεγόμενος ε, επανορθωτικός γάμος. Η δε δολοφονία της ε, συζύγου τιμωρούνταν ε, με επίοικια αν ο σύζυγος θεωρούσε ότι υπάρχει μοιχεία. Η δε, ο δε βιασμός μέχρι το 1994 δεν ήταν ένα έγκλημα κατά συγκεκριμένου προσώπου, αλλά κατά των χριστών ηθών και μόνο έξι μήνες μετά το συμβάν μπορούσε η γυναίκα να το καταγγείλει. Μετά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή είναι σαν να έχει γραφτεί ο νόμος για να μην υπάρχει δίωξη του βιασμού. Να παριστάνουμε ότι δεν συμβαίνει καν. Ένας νόμος που έχει γραφτεί από άντρε για άντρε. Για να προστατεύει τους βιαστές. Με βίασαν το 97. Χρειάστηκαν 20 χρόνια για να το επεξεργαστώ μέσα μου να βρω το κουράγιο για να μιλήσω δημοσίως. Και δεν ε, έλαβε καν χώρα στην ε, Ιταλία, αλλά στην Γαλλία. Τι πιθανότητες είχα 22 ετών να ε, βρω δικαιοσύνη. Όχι να με πιστέψει μόνο η κοινή γνώμη, αλλά και το δικαστήριο απέναντι σε έναν από τους πιο ισχυρούς παραγωγούς του Hollywood. Γνωρίζοντα ότι απέναντί μου είχαν έναν άντρα στην κορφή της πυραμίδας εξουσίας ο οποίος θα κατέστρεφε οποιαδήποτε καριέρα είχα. Τα χέρια μου ήταν δεμένα και το στόμα μου κλεισμένο. Και δεν ήμουν η μόνη. Δεκάδες γυναίκες ε, είχαν ε, υποστεί επιθέσεις από τον ίδιο άντρα και σιωπούσαν γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή. Γιατί οι καριέρες μας πεζότανα. και μάλιστα είχαμε υπογράψει και συμφωνίες εμπιστευτικότητας που έλεγαν ότι θα υποστούμε οικονομική καταστροφή αν μιλούσαμε ποτέ. Με το πιστόλι στον κρόταφο δηλαδή συγκαλύπταμε τον ίδιο μας το βιασμό. Ζούσαμε σε καθεστώς φόβου και παράνοιας. Κάποιες διαπιστώσαμε αργότερα ότι μας παρακολουθούσαν και μας φακέλωναν την ιδιωτική μας ε, ζωή, οποιαδήποτε διακρισία μικρή ή μεγάλη, έτοιμη φάκελοι για να μας καταστρέψουν ανα πάσα στιγμή. Όταν τελικά αποφάσισα να μιλήσω, στην Ιταλία δεν πίστεψαν την ε, <coughs> πτωσή μου. Ήδη με θεωρούσαν πόρνη εκεί. Η ιστορία δε αυτή θεωρούσαν ότι ήταν η επιβεβαίωση. Έσυρε το όνομά μου στην λάσπη και η υπόλοιψή μου σπηλώθηκε. Η αξιοπιστία μου αμφισβητήθηκε. Κάθε μέρα στην τηλεόραση γινόταν μια συζήτηση από ανθρώπους που δεν με ήξεραν, τους οποίους δεν έχω συναντήσει ποτέ μου και συζητούσαν αν με βίασε ή όχι. Συζητούσαν για τη ζωή μου σαν να ήταν detective σε κάποια σκηνή εγκλήματος που υπήρχε μόνο στην ε, φαντασία τους. Όλα αυτά σε κάθε κανάλι την ώρα εχνής και το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι το ήθελα κιόλας. Όχι ότι το άξιζα μόνο. Δηλαδή δεν ήμουν, ε, δεν μου άξιζε καν ο βιασμός. Μετά από αυτή την ε, δαιμονοποίησή μου και αφού ξαναζούσα το δράμα μου και το τραύμα μου δημοσίως έπεσα σε βαθιά κατάθλιψη για μήνες. Η πιο βαριά κατάθλιψη που είχα ζήσει ποτέ. Και κατάφερα να το ξεπεράσω μόνο χάρη στην απίστευτη στήριξη των δύο δύο οργανώσεων των φεμινιστικών της ε, Ιταλίας που με στήριξαν. Και βεβαίως ε, και των φίλων μου Ροζ Μαγκάουαν, Ροζάνα Αργέτ, ε, των υπολείπων θυμάτων αυτού του ανθρώπου. Και τελικά σταθήκαμε ενωμένε και πιο δυνατές. Και σε όλη αυτή την δοκιμασία μεταμορφώθηκα. Τελικά είχα ένα ρόλο που δεν είχα σκεφτεί ποτέ να αναλάβω, αλλά τελικά δεν είχα καμία επιλογή παρά να παίξω αυτών τη ακτιβίστριας. Ε, Έπρεπε να μιλήσει για τι γυναίκε που δεν είχαν βρει το φάρος ακόμα να μιλήσουν και να ακουστούν και τώρα. Ελπίζω και πιστεύω ότι λόγω του μύτου, αυτού του παγκοσμίου φαινομένου στα κοινωνικά μέσα, ότι κάθε γυναίκα έχει φωνή, έχει την ευκαιρία να μιλήσει και θα είμαστε ενωμένε. Οι φωνές μας ε, μαζί θα γίνουν βρυχυθμός και έτσι θα υψώσουμε την φωνή της αγανάκτησής μας και επιτέλους μας ακούν και μας πιστεύουν. Αυτό το μη θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα να είναι η μεγαλύτερη επανάσταση που έχει γίνει για τις γυναίκες από το δικαίωμα ψήφου. Μια πορεία προς την ισότητα για την δικαιοσύνη και έχω την τιμή να είμαι ένα μικρό μέρος του και να σας μιλάω σήμερα. Όταν ήμουν μικρό κοριτσάκι και έπαιζα στις ταινίες, Ποτέ δεν ονειρευόμουν ότι θα με ακούσει κάποιος. Πώς θα φανταζόμουν ότι μια μέρα θα μιλούσα για τη ζωή μου, για το τραύμα μου, για την επιβίωσή μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αύριο στις 8 Μαρτίου στους δρόμους της ε, Ρώμης ε, θα βαδίσω μαζί με τις ε, υπόλοιπες γυναίκες ακριβώς που έχουμε την ίδια εμπειρία. Δεν είμαστε πια θύματα νικάμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε από εμάς, ανά πάσα στιγμή. Ναι, πράγματι. Γιατί? Γιατί λόγω της ε, ισορροπίας εξουσιών, λόγω της κατάχρησης εξουσίας, γιατί οι άνδρες έχουν την εξουσία σχεδόν παντού. Και μέχρι σήμερα η φωνή μας δεν ακουγόταν. Θα μπορούσα να είμαι εγώ, εσείς, η κόρη μου, η μητέρα μου. Πολλές από εμάς ε, πιθανότητα να έχουμε μια παρόμοια εμπειρία και απλά θέλησαμε να την ξεχάσουμε ή δεν θέλησαμε να συμβιβαστούμε. Όπως και εγώ, οι αδελφές μας, οι φίλες μας. Έτσι λοιπόν. Πόσο βέβαια είστε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν με αυτή τη δράση. Θα είδατε τα Όσκαρ της προάλλες. Δεν με ενδιαφέρουν τα Όσκαρ. Ναι, συγκινούμε βέβαια που οι άνθρωποι αναγκάζονται σήμερα να συζητήσουν τα θέματα αυτά αφού τόσες πολλές ηθοποιοί και άνθρωποι που εργάζονται βιομηχανία του κινηματογράφου εκφράζονται ελεύθερα και φυσικά αν δεν μιλούσαν τα Όσκαρ θα τα κατηγορούσαν ως υποκριτικά, κάτι που για μένα είναι προφανές. Ε, δεν ανήκω στο Hollywood, οπότε δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Καλό είναι που ε, αναφέρουν τα θύματα που γυναίκες που καταστράφηκαν οι καριέρα τους, η καριέρα τους από αυτό το τέρας. Πώς βλέπετε να τελειώνει, ποιο θα είναι το τέλος του τέρατος. Θα ήθελα να μπορώ να πω ότι αυτό το τέρας και τα άλλα τέρατα που εγώ χρειάστηκε να συναντήσω θα καταστραφούν από τις γυναίκες και τους άντρες που αυτοί βίασαν, αλλά δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα είναι η δική μας γενιά. Όπως ο Αλκαπόνο δεν θα είναι, ούτε όπως η φοροδιαφυγή, όπως τα άλλα ζητήματα. Έχω αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε εμείς αυτή την ευκαιρία στη ζωή μας αλλά είμαι βέβαιη ότι όχι λόγω κάρμα μόνο, αλλά ότι με κάποιον τρόπο θα το πληρώσει. Θέλω να σας ζητήσω το απίστευτο, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Το αδιανόητο θα σας ρωτήσω. Έχουν γίνει έρευνες στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ένας γιατρός ε, εκτακτών περιστατικών που μίλησε σε μια κλινική για θύματα ε, με, με εγκαυμάτων ότι λέει ότι έχει δει σωματικά αποτελέσματα, θεραπεία τα οποία εμφανίζονται όταν φτάνει κάποιος στη στιγμή όπου πρώτα συγχωρεί δηλαδή ότι σε ένα πεντάλεπτο αρχίζει μια συζήτηση με το θύμα και τους ζητά να συγχωρέσουν τον εαυτό τους τον εγκληματία, το, το, το πεζοδρόμιο που κάτι έγινε. Κοιτάξτε, ναι, μπορεί να το πει όπως θέλει κανείς, χριστιανικό, πνευματικό, αλλά εγώ θέλω δικαιοσύνη και τη δικαιοσύνη τη φτιάχνουν οι άνθρωποι, όχι ο Θεός εδώ πάνω στη γη. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτοί. Αν τον συγχωρώ καθόλου, ποτέ θα θεραπευθώ μια χαρά με την ε, δύναμή μου, με τη δύναμη των άλλων γυναικών, με τον βρυχηθμό μας, με την εκδίκησή μας, με την ε, επανάστασή μας, με το κίνημά μας. Αυτό θα είναι η θεραπεία μου, όχι με τη συγχώρεση. Αυτά να τα συνεννοηθεί αυτός με το δικό του Θεό, όχι με το δικό μου. Θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις, παρακαλώ. Μην είστε δειλές, κάντε μου ερωτήσεις. Έχουν μείνει αποσβολωμένε. Γεια σας, λέγομαι Θερίσα Κίσλερ, είμαι Σουηδή δημοσιογράφος. Φρικτή αυτή η μεταχείριση που συζητήθηκε για αυτή την κατάσταση της Ιταλίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν περάσει χρόνια. Υπάρχει κάποια αυτοκριτική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ιταλία μετά από όλα αυτά. Είναι λιγότερο από ένα χρόνο. Είναι από τον Οκτώβριο. Αφού έγραψαν άρθρα παγκοσμίω για την εσχρή μισογενιστική μας ε, ε, πατριαρχική κοινωνία στην Ιταλία και για τα μέσα μας που λειτουργούν αντίστοιχα και για τα θύματα, τότε άρχισαν να σταματούν σιγά σιγά να ντροπιάζουν τα θύματα. Αφού δηλαδή όλος ο υπόλοιπος κόσμος έγραψε εκτενή άρθρα κατανομάζοντας τις εφημερίδες τους, τους δημοσιογράφους αυτούς, το τι είπαν, γιατί αυτό σοκάρισε τον υπόλοιπο κόσμο, το ότι πήγαν να το αποσιωπήσουν, παρότι μερικοί συνέχισαν. Ακόμη και εγώ σήμερα για αυτούς αποτελούν ντροπή. Είναι κάτι που σίγουρα θα μετανιώσουν αύριο και εγώ δεν δίνω δεκάρο. Μια ερώτηση. Από τη Γερμανία προέρχομαι εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω, σκέφτεστε μήπως να γράψετε κάποιο βιβλίο? Έκανα μία ταινία, είναι απάντηση, για το βιασμό μου. Ενάμιση χρόνο μετά το βιασμό. Οπότε την κάθαρσή μου την έκανα τότε. Για να το ξεπεράσω, παρόλο που δεν το ξεπέρασα. Και ήταν και είναι η μόνη απόδειξη που έχω. Γιατί δεν το ήξερα, αλλά ακριβώς εκεί περιέγραψα σε αυτή την ταινία το modus operandi. Πώς δηλαδή το κάνει, ότι σε εκπλήσει, έρχεται με το μπουρνούζι του, σου ζητάει μασάζ, Κανένα τότε το 99 που το, το έφτιαξε αυτό, έφτιαξε αυτή την ταινία, δεν το πίστευσε. Δεν ξέρω αν ε, μπορεί να βοηθήσει στο να γεμίσει το πάζλ, να φτιαχτεί. Ένα βιβλίο. Όχι με τη δική μου φωνή, δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαι μόνη μου. Ήμουνα μόνη μου μια ζωή. Θεωρώ ότι είμαι μέρος μιας ομάδας και θέλω να παραμείνω μέλος αυτής της ομάδας που με βοήθησε να αποφύγω αυτόν τον ε, αποκλεισμό τελικά, να το σταματήσω. Οπότε αν υπάρξει ένα βιβλίο θα προτιμούσα να το γράψουμε πολλές μαζί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτή την ε, ταινία, όχι «Ε, τίποτα μακάβριο. Κάτι το οποίο με εκπλήσει είναι ιστορίες για ε, σεξουαλική βία σε βάρος ε, γυναικών και πώς ε, μετά αυτό διονύζεται μερικές φορές. Εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα, να δώσω παραδείγματα, αλλά μερικές φορές βλέπουμε να διονύζεται μια ιστορία, τα βλέπουμε αυτά σε ταινίες δηλαδή, έτσι, ότι όταν κάποιος έχει υποστεί σεξουαλική βία, στη συνέχεια και ο ίδιος προβαίνει σε σεξουαλική βία, ίσως 20 χρόνια αργότερα. Ναι, ναι, όντως, και το είπα κιόλα. Όντως, φτάνουμε να κάνουμε ακραία πράγματα. Δηλαδή, ναι, λέμε μια ιστορία. Η ταινία αυτή είναι μια ταινία, έτσι. Υπάρχει κάμερα, υπάρχει κόσμος γύρω. Έχει αποδειχτεί ότι οι ηθοποιοί σε μια σκηνή που τσακώνονται, αυτό που συμβαίνει μέσα στον οργανισμό τους είναι το ίδιο που συμβαίνει όταν έχουν μια πραγματική μάχη με κάποιον, όταν τσακώνονται πραγματικά με κάποιον. Δηλαδή είναι πολύ λεπτή γραμμή διαχωρισμού. Και εδώ, ξέρετε, δεν είμαι πραγματικά εθοποιος τώρα, το 2013 σταμάτησα. Τώρα, σκηνοθετώ, όταν κάποιος ε, σκηνοθετεί, βρίσκεται σε μια πιο έτσι ήπια κατάσταση. Η ιεραρχία, η πυραμίδα είναι λιγότερο απόλυτη και αυστηρή. Πρόκειται περισσότερο για συνεργασία. Οπότε δεν ταυτίζομαι πια με την ηθοποία. Μπορώ να σας πω ότι πάντα ντρεπόμουν στη ζωή μου που ήμουν ηθοποιός, δεν ξέρω γιατί. Και αισθάνεστε τι, όπως όταν ετοιμάζεται κανείς να πάει στο χορό και ρουφάει την κοιλιά του και δεν τον κορσέ και ετοιμάζεται να βάλει. Η Μέρη Στριπ, για παράδειγμα, πληρώνει για να... Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τη Μέρι Στριπ. Ωραία, πείτε μας το δικό σας το αφήγημα. Αναφερθήκατε στη θυματοποίηση. Τώρα βάζουμε λέξεις στο φαινόμενο το Mansplain για παράδειγμα που είπαμε πριν, ε, ξαφνικά εμφανίζονται καινούργιες λέξεις, καινούργια ορολογία για να περιγράψουμε κάτι που παλιά δυσκολευόμασταν, σαν ασθενογραφία. Οι λέξεις έχουν σημασία. Με ελευθερώνουν οι λέξεις που βγαίνουν από το στόμα μου, πράγματι. Έπειτα είμαστε σε ένα νέο κόσμο πια. Σε ένα κόσμο που θα πετύχουμε την ισότητα αντρών και γυναικών για τις κόρες μας, για τις επόμενες γενιές. Κάτι έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό. Πια δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτό το κίνημα, δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Θα πρέπει να τα καταφέρουμε, γιατί αν χάσουμε αυτή τη στιγμή, η συζήτηση γίνεται όλο και περισσότερο. Αποκτά διαστάσεις. Οπότε και σε εσά ζητάω να συνεχίσετε να το συζητάτε, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και σπίτι σας, με τους φίλους σας. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και πρέπει να συνεχίσει το είδο μας με ισότητα μεταξύ των δύο φίλων και εγώ να ρωτήσω κατά πόσο εσείς διώξατε τα μέσα ενημέρωση στην Ιταλία για δεσφήμιση. Και τι πρέπει να κάνουμε με αυτή την οτροπία την σεξιστική που εμφανίζει τη γυναίκα πάντα σαν ε, σεξουαλικό αντικείμενο. Κοιτάξτε. Ναι, όντως πήγα στη δικαιοσύνη για διάφορους εφημερίδες, Όντω. Θα μπορούσα ε, να φτάσω για 12 περιπτώσει στα δικαστήρια, αλλά αυτό κόστιζε ακριβά. Οπότε ζήτησα από φεμινιστικέ ε, οργανώσεις να με βοηθήσουν, πήρα ένα δικηγόρο, πήγα στη δικαιοσύνη και κέρδισα. Και τα χρήματα αυτά θα πάνε σε ανεξάρτητε φεμινιστικέ ομάδες και οργανώσεις, το Κάζα Ντελαντόνα στη Ρώμη για παράδειγμα που κινδυνεύει να κλείσει. Τι πρέπει να κάνουμε για το σεξισμό στα, στις ταινίε. Εγώ σκέφτομαι τώρα τι πρέπει να κάνουμε για να συνεχιστεί αυτό το κίνημα. Γιατί αν συνεχίσουμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα, θα αλλάξει και ο τρόπος που γίνονται οι ταινίες θα γίνονται με διαφορετική οπτική. Αν έχουμε περισσότερες γυναίκες σκηνοθέτηδες, αν έχουμε περισσότερες γυναίκες συγγραφείς, θα παρουσιαστεί μια διαφορετική οπτική. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ωραία τελικά, χρήματα μπαίνουν στην πάντα για νομική στήριξη. Δεν θέλω να μπω σε αυτό, ναι, είναι πολύ Hollywood αυτό. Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του Ταμείου κανένα θύμα, καμία από εμά που διακινδυνεύουμε τα πάντα. Όταν εγώ πρωτομίλησα, σας είπα, ήμουν η πρώτη που μίλησε, η πρώτη που έδωσε πληροφορίες. Εντάξει, όχι η πρώτη που μίλησα μάλλον, να το πω πιο σωστά, αλλά η πρώτη που κατέγραψε το αφήγημά της. εξαναγκάστηκα λίγο πολύ και το είπα. Να τη ιστορία μου, να το όνομά μου, πείτε το και στις άλλες γυναίκες, δεν ξέρω τα ονόματά τους, αλλά να τους το πείτε ότι εγώ θα δημοσιοποιήσω την ιστορία μου. Και ευτυχώς εμφανίστηκε η γυναικεία αλληλεγγύη. Ήτανε τεράστια. Τόσες άλλες γυναίκες που διακινδύνευσε και αυτές πηγαίνοντας ενάντια στον πιο ισχυρό άνθρωπο του Χόλιγουτ που ε, με τη σειρά του πήγε στη δικαιοσύνη του New York Times. Αλλά βέβαια μετά τόσο πολλοί κόσμος που βγήκε η πραγματική ιστορία. Διακινδυνεύουμε πολλά. Η οργή ήταν τόσο μεγάλη, ούτε και εγώ κατάλαβα ότι ήταν τόσο πολλές οι γυναίκες θύματα, αποφάσισα ότι είμαι έτοιμη να τα διακινδυνεύσω όλα. Όταν βλέπουμε πόσοι είναι εναντίον μας και πόσοι ήταν έτοιμοι να μας καταδικάσουν και αυτός ο άνθρωπος, βλέπετε, εξακολουθεί να βρίσκεται ελεύθερος. Σε ένα σπά στην Αριζόνα βρίσκεται σε μια κλινική για ε, εθισμό στο σεξ. Μα τι λέμε τώρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν θέμα εθισμού. Είναι ψυχοπαθής. Το θέμα είναι να δείχνει κανείς ότι συμπάσχει με τους άλλους. Γι' αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει θεραπεία, όπως για τους serial killers. Πως πρέπει να σταματήσουμε να επιβραβεύουμε τη συμπεριφορά των ψυχοπαθών που διακρίνουμε στους ηγέτες μας. Εσείς είπατε τη δικιά σας ιστορία. Ας δούμε όμως και άλλες ιστορίες σε άλλους κλάδους, στην πολιτική ιδιαίτερα. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπουμε, για τον Τραμπ, συγγνώμη που το λέω εντάξει είναι κάτι που εμένα προσωπικά με απασχολεί. Εμφανίστηκε πλήρως διαμορφωμένος Δεν ήταν μια τάση που πέρασε και στην επόμενη γενιά όλα θα είναι ωραία και καλά. Όχι. Υπάρχουν αυτά τα μεγάλα σκοτεινά τέρατα και γι' αυτό ρωτάω, όχι για το συγκεκριμένο τέρας, αλλά για τα τέρατα που υπάρχουν παντού στο είδος μας. Πώς σκοτώνουμε τέτοιου είδους τέρατα. Ε, το να σκοτώσουμε είναι έγκλημα, έτσι. Ναι, ενώ ψυχολογικά το φόνο, έτσι. Ναι, πρέπει να υψώσουμε τη φωνή μας και να δείξουμε αλληλεγγύη απέναντι στις γυναίκες. Να μην αμφιβάλλουμε όταν έρχονται οι γυναίκες και διηγούνται αυτές τις ιστορίες, γιατί αν δεν πιστέψουμε τις άλλες ιστορίες, τότε ποιος θα μας πιστέψει εμάς. Εμείς οι γυναίκες λοιπόν όταν μιλάμε για αυτούς που μας βίασαν έχουμε να χάσουμε τα πάντα. Εγώ όμως δεν ήθελα χρήματα. Επέλεξα να βγω και να τα πω. Άρα αυτό που είναι να με πιστέψουν. Να πιστεύουμε τις γυναίκες. Να φωνάξουμε. Δεν πειράζει. Ας εξοργιστούμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε το τέλειο θύμα. Ας υπάρχουν και οργισμένα θύματα. Γιατί όχι. Και εγώ με τις αδερφές μου τσακώνομαι, με δημοσιογράφους μερικές φορές. Δεν πειράζει. Και εμείς έχουμε το δικαίωμα να φωνάξουμε και να τσακωθούμε μερικές φορές. Γιατί όχι. Συγγνώμη, εσείς πήρατε το λόγο ήδη μια φορά. Παρακαλώ, εσείς. Η Λίεβα από το περιοδικό ΕΒΑ της Βουλγαρίας. Είσαστε πολύ θαραλέα. Γι' αυτό που κάνατε νομίζω ότι δεν αλλάζετε μόνο τον εαυτό σας αλλά και την κοινωνία. Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, με τα παιδιά σας το έχετε συζητήσει. Και ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για σας να μιλήσετε με αυτά. Όσον αφορά τα παιδιά μου, έχω μια κόρη 16χρονη. Τη είπα, πριν τη είχα πει ότι κάτι είχε συμβεί σε μένα. Δεν τη είπα τις λεπτομέρειες, αλλά ήθελα να ξέρει ότι κάτι υπήρχε. Μετά αναγκάστηκα. Ούτε στον πατέρα μου το είχα πει. Πριν λίγες μέρες πριν βγω να τα πω ε, έξω τα είπα και αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα γι' αυτόν. Ήξερα ότι θα πληγωθεί και στο γιο μου. Ένα χρόνο ήταν πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολύ προσωπικό όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο. Ούτε για μένα ούτε για την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και τους αγαπημένους μου. το τραύμα που έζησα εγώ το πέρασα και σε άλλους. Επειδή ακριβώς εγώ το έζησα. Και το άλλο που με ρωτήσατε, το μεγαλύτερο φόβο σας όταν τα διηγήθηκατε όλα αυτά. Ναι, ήταν ένα άλμα στο κενό. Δεν ήξερα τι να περιμένω. Δεν περίμενα ότι κάποιος θα στραφεί εναντίον μου ή τέλος πάντων, ωραία, το είχα υποθέσει, δεν ήταν αυτό το φόβος μου ακριβώ. αλλά ήταν ακριβώς αυτό, άλμα στο κενό. Έγιναν τα πράγματα τόσο γρήγορα, μέσα σε μια εβδομάδα δεν είχα καιρό να φοβηθώ. Όμως από τη στιγμή που άρχισα να μιλάω γι' αυτό και είπα το όνομά μου, βγήκε το πρώτο άρθρο, σε δέκα μέρες γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβα να φοβηθώ. Σαν πύραυλος. Εκτοξεύθηκα σε αυτήν την αποκάλυψη. Βγήκα με αυτήν την αδιαφυσβήτητη αλήθεια που έπρεπε να βγει, ήταν πιο δυνατό από μένα. Ευτυχώς. Ναι, τώρα λέω και εγώ ευτυχώς. Ευτυχώς, ναι. Παρακαλώ. Ε, Μαρία Χούκλη από Αθήνα 984 και Inside Story από την Ελλάδα. Ε, Κυρία Argento, no? No, no, Greece. Sorry, I can't quite hear you. yes. Πραγματικά, μπράβο σας για το θάρρος που βρήκατε να... so many languages. quickly. Μπράβο για το θάρρος που βρήκατε. Can you hear me? No? I don't hear the... It's coming. English. There, there. Okay, right? italiano. Okay. Λέω μπράβο για το θάρρος που βρήκατε να δημοσιοποιήσετε αυτή την τραγική περιπέτειά σας, αυτόν τον εφιάλτη. Νωρίτερα είπατε ότι οι γυναίκες πρέπει να πιστεύουμε τις γυναίκες και να τις στηρίζουμε. Θα γνωρίζετε προφανώς ότι έχει ασκηθεί κριτική στο κίνημα MeToo από επιφανείς γυναίκες όπως η Κατρίν Ντονεύ και άλλες ε, οι οποίες θεωρούν ότι οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση φτάνουν στο άλλο άκρο και ουσιαστικά οδηγούν σε μια πολιτική ορθότητα που καταδικάζει και τις σχέσεις ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών, το φλερτ, ε, ότι έχει φτάσει στα άκρα δηλαδή ε, να διαχωρίσει τα δύο φύλλα. Θα προσθέσω και ένα ακόμη ερώτημα γιατί εσείς διαχωρίσατε τη θέση σας από το μανιφέστο των Ιταλίδων που κατήγγυλαν τη σεξουαλική παρενόχληση χωρίς βεβαίως να καταγγελούν συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά στάθηκαν στο πλευρό του κινήματος μήτου Αυτά τα δύο ερωτήματα. Mm, yes. Okay. Ναι, μάλιστα. Ε, νομίζω ότι είναι σαφές για τις ε, γυναίκες ε, το τι εστί παρενόχληση, βιασμός, κακοποίηση και το τι είναι φλερτ ε, και καμάκι. Έτσι δεν υπάρχει, δεν είναι γκρίζα η γραμμή, είναι σαφές. Θέλω να φλερτάρω, θέλεις να φλερτάρεις, το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι... Η φίλη μου, η Ρόζ Μαγκάμαν, μου είπε, είπε κάτι και συμφωνώ πλήρω. Αν η Κατρίν Τενεύ και ίσω οι γυναίκε αυτή τη γενιά που υπέγραψαν αυτή την επιστολή ε, μπορούσαν να δουν πόσε φορέ ε, στην ε, ζωή τους πέρασαν το ίδιο πράγμα, ταπεινώθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν και κακοποιήθηκαν, θα είχαν ε, τρελαθεί. Οπότε είναι ευκολότερο να το αποφύγουν τελείως και συμφωνώ με τη Ρόζ. Όσον αφορά τώρα το τι ακριβώς ε, έγινε στην Ιταλία, καμία από αυτές ε, τις Ιταλίδες που υπέγραψαν αυτή την έκκληση στην κοινή λογική δεν μου έγραψαν, ε, δεν ήρθαν σε επαφή μαζί μου, δεν με πήραν τηλέφωνο, δεν είχαν πει τίποτα. Επί πέντε μήνες έγραψαν ένα μανιφέστο χωρίς να έρθουν σε επαφή μαζί μου. Ε, ήρθαν με ένα κείμενο έτοιμο, γραμμένο, ε, δεν κατονόμαζαν εμένα ή την άλλη Ιταλίδα που μίλησε, η Μυριάννα Τρεβιζάνη ή την... και η Άμπρα Μπατιλάνο. Όχι μιλούσαν για γενναίες γυναίκες ε, γυναικός. Ε. Εντάξει δεν κρατάω κακές, αλλά είναι αυτό πολύ λίγο που έγινε και πολύ αργά. Και εγώ δεν αισθάνομαι μέλος αυτής της ομάδας, ε, δεν με περιέλαβαν. Μου ζήτησαν να υπογράψω ένα γράμμα. Εγώ, δηλαδή εντάξει, εγώ ήμουνα στα χαρακόμματα επί μήνες και τώρα μου λέτε έλα να, να υπογράψεις. Και λέμε και λένε κιόλα δεν δείχνουμε τον συγκεκριμένο με το δάχτυλο, αλλά γενικώ όσου κακοποιούν και το σύστημα. Μα δεν πάει έτσι, δεν, θα κερδίσουμε έτσι τον πόλεμο. Με το να λέμε με κακοποίησε ο Χίψη και τα λοιπά. Έτσι θα το κάνουμε. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι το έκαναν για να καθισχάσουν τη συνείδησή τους για την εκοφαντική σιωπή. Τελεία και Παύλα. Και μας συγχωρείτε οι ερμηνείς ε, ξεπέρασαν και το ωράριό τους γιατί άξιζε βεβαίως να ακουστεί αυτή η ιστορία σε όλες τις γλώσσες. Σας ευχαριστούμε. Ε, ευχαριστώ και σας για την συζήτηση αυτή, για τις δύσκολες ερωτήσεις. Έχω πολύ ύλη να γράψω φοβερές ιστορίες ε, μεταξύ των οποίων και αυτή η συγκλονιστική ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι ο εαυτός μου, μια γυναίκα.